Bonjour à toutes et à tous. Καλημέρα. Και πάλι θα αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας χωρίς άλλη καθυστέρηση, διότι είναι μεγάλο προνόμιο για μας που μπορούμε να υποδεχτούμε εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, αυτήν την ε, κοινή επιτροπή με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην συζήτηση που θα έχουμε για τη Συρία. Θα συζητήσουμε εδώ την κατάσταση στη Συρία και τις επιπτώσεις που έχει σε όλη την γύρω περιοχή. Η κατάσταση επιτόπου, όλοι το γνωρίζουμε, είναι τραγική και δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς πως μπορεί να χειροτερέψει περισσότερο. Ιδίως μάλιστα τώρα που φτάνει ο χειμώνας και η βία συνεχίζεται. Πάνω από 2.200.000 πρόσφυγες έχουν μαζευτεί. Πολλοί από αυτούς είναι παιδιά, μια χαμένη γενιά δηλαδή. Οι γείτονε χώρε προς τη Συρία πρέπει και αυτές να αντέξουν ένα όλο και μεγαλύτερο βάρος, αφού πρέπει να υποδεχτούν όλο και περισσότερους μετανάστες, πρόσφυγες μάλλον. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να προσφέρει όλη τη βοήθεια που μπορεί για να παραμείνουν τα σύνορα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της είναι οι πιο σημαντικοί δωρητές στην περιοχή. Είναι αυτοί που έχουν δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Ένα ποσό το οποίο σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Χιωρίλα Προβέρα, εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ιδιαιτερότητε τη κρίση στη Συρία και οι συνέπειέ τη στι κοινωνικέ, πολιτικέ και οικονομικέ δομέ τη χώρα απαιτούν από πλευρά μα μία παρέμβαση διαρκή, μακροπρόθεσμη, συνολική, διεθνούς χαρακτήρα που να μην αντιμετωπίζει μόνο την κατεπίγουσα ανθρωπιστική κατάσταση. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την πολιτική μας και διπλωματική μας δράση προκειμένου να σταθεροποιηθεί ολόκληρη η γεωγραφική αυτή ζώνη. Επίσης να καλύψουμε όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και μειονότητες που πλήττονται από αυτή τη σύραξη και που στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουν την ανοικοδόμηση της χώρας. Αυτός ο διεθνής συντονισμός απαιτείται για να υλοποιηθούν συγκεκριμένα και κοινά προγράμματα ώστε να μπορέσει μια μέρα να φτιαχτεί ξανά το μέλλον της Συρίας και να σταθεροποιηθούν οι χώρες της περιοχής που έχουν υποδεχτεί τόσες χιλιάδες πρόσφυγες. Η ανάγκη αυτής της διεθνούς παρέμβασης επιβεβαιώνεται από την παρουσία των επιτροπών, των ε, κυρίων φορέων του ΟΗΕ που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, ώστε να συζητήσουν μαζί μας τις ενδεχόμενες νέες στρατηγικές βοήθειας προς τη Συρία και τις γείτονες χώρες της. Μην ξεχνούμε ότι η λύση στην κρίση της Συρίας πρέπει πάνω απ' όλα να είναι πολιτικού χαρακτήρα. Α, έτσι είναι εύστοχη η παρουσία του Γενικού Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, του κ. Ντιμό, τον οποίο χαιρετώ, και ο οποίο μόλι έφτασε από τη Γενέβη. Ο κύριος Βιλμό θα μπορεί να μας ενημερώσει για το τι συνέβη στη συνεδρίαση της Γενέβης 2. Πριν δώσω το λόγο επίσης στην Επίτροπο Γεωργίευα για το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης, κοινή συνεδρίασης με τους βασικούς διεθνείς φορείς για τη βοήθεια προς τη Συρία, θα ήθελα εξ ονόματος όλων να κάνω έκκληση ζητώντας την απελευθέρωση της κυρίας Ραζάν Ζαϊτουνέ, βραβείο ε, που έχει κερδίσει το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία απήχθη στη Συρία ε, μαζί με τον σύζυγό τη και τη οποία αγνοούμε την τύχη. Να περάσουμε τώρα στι παρεμβάσει των προσκεκλημένων μα, που θα ζητήσω να είναι συνοπτικοί στι ομιλίε του, ώστε να έχουμε μετά πολύ χρόνο για συζήτηση και ρώτα απαντήσει με του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Να ευχαριστήσω του δύο συμπρόεδρους στη συνεδρίαση αυτή, αλλά να ευχαριστήσω και το καθένα από τους ευρωβουλευτές που μας στήριξαν κατά τη διάρκεια των χιλίων ημερών σύραξη στη Συρία, που μας στήριξαν στο έργο μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν υποφέρει τόσο πολύ μέσα στην ίδια τη χώρα αλλά και στις γείτονες χώρες. Η κρίση αυτή είναι ιδιαίτερη. Μας αγγίζει όλους. Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για Σύριους οι οποίοι μάχονται ο ένας τον άλλον είναι κάτι που έχουμε στη συνείδησή μας όλοι, διότι δεν καταφέρνουμε να βρούμε έναν τρόπο να πιέσουμε τις διάφορες πλευρές της σύγκρουσης αυτής, ώστε να σταματήσει για να σωθούν οι άνθρωποι, για να προστατευτεί η περιοχή και να υπάρξει σταθερότητα. 22 Ιανουαρίου Ελπίζουμε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και εμείς από την ανθρωπιστική κοινότητα ευχόμαστε οι διαπραγματεύσεις αυτές να οδηγήσουν στην ειρήνη. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η μιζέρια που πλήττει το λαό της Συρίας. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης για μια σημαντική συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί με τους επικεφαλείς των ανθρωπιστικών ε, υπηρεσιών του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την Διεθνή Τράπεζα και τους δωρητές που στηρίζουν τους ίδιους. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρία θέματα. Πρώτον, μια συνολική απάντηση στην κρίση. Συνολική με την έννοια ότι έχει ως στόχο την Συρία και τις γείτονες χώρες. Θέλουμε δηλαδή να προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες, αλλά να προσφέρουμε και μακροοικονομική στήριξη, ιδιαίτερα στην Ιορδανία και το Λίβανο. Έχουμε ακολουθήσει έναν μακρύ δρόμο για να πείσουμε την ανθρωπιστική κοινότητα να συνεργαστεί έτσι ώστε να υπάρξει μαζική στήριξη για να σωθούν οι ζωές αλλά και για να υπάρξει σταθεροποίηση στην περιοχή. Εδώ θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αυριξιακή βοήθεια που προσέφεραν διάφορες οργανώσεις, ώστε να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε μια ολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης στον ανθρωπιστικό τομέα. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στους Ευρωπαίους, γιατί οι Ευρωπαίοι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το είδαμε και είπαμε από την αρχή ότι στην κρίση αυτή εξαιτίας της φύσης της και εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει σε ολόκληρη την περιοχή δεν φτάνει η συνηθισμένη ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες και στις γείτονες χώρες. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της χρηματοδότησης. Τα Ηνωμένα Έθνη ήρθαν με τη μεγαλύτερη δυνατόν ποτέ έκκληση τη Δευτέρα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια για δράση μέσα στη Συρία αλλά και στις γείτονες χώρες. Η έκκληση αυτή αντικατοπτρίζει τη θλιβερή πραγματικότητα των αναγκών που όλο και αυξάνονται στη Συρία και στην περιοχή. Ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια μέσα στη Συρία τώρα είναι περίπου 10 εκατομμύρια, 9,3. Οι μετατοπισμένοι μέσα στη χώρα είναι 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι μετατοπισμένοι στις γείτονε χώρες είναι 2,3 εκατομμύρια. Και γνωρίζουμε και το βλέπετε κι εσείς στις ειδήσει, στην τηλεόραση, τι συμβαίνει με το χειμώνα. είναι ένας πληθυσμός που συνήθως δεν είναι συνηθισμένοι σε πολύ σκληρούς χειμώνες όπως έχουν φέτος, δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν πρόσβαση γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Συρία, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που γίνονται μάχες, το να δίνει κανείς λεφτά δεν κάνει διαφορά, γιατί πρέπει να φτάσουμε για να τους προσφέρουμε βοήθεια ή να τους δώσουμε την ευκαιρία να φύγουν από τις περιοχές αυτές ή και τα δύο βέβαια. Οπότε για το θέμα αυτό της πρόσβασης ακούσαμε και από τον Πέτερ Μάριουμ και από διάφορες οργανώσεις και από τον Κουζέν ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει πολιτική δέσμευση όποιος μπορεί να μιλήσει με τις πλευρές που συμμετέχουν στη σύγκρουση αυτή να το κάνει για να τους πείσει να βοηθήσουν να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών δεν φτάνει μόνο με το ψήφισμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στη συνάντηση αυτή λοιπόν σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε και με τα παιδιά στη Συρία που είναι τα πιο ευάλωτα. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τον Λίκη για τη δουλειά που έκανε από πλευρά της UNICEF για να πλαισιώσει ένα πρόγραμμα για την γενιά αυτή, ένα οριζόντιο πρόγραμμα μέσα στη Συρία για να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, εμβόλια κατά της πολιομελίτιδας και άλλων ασθενειών σε συνεργασία με άλλες χώρες που μπορούν να δεχτούν πρόσφυγες παιδιά ώστε να μπορούν αυτά να πάνε στο σχολείο και γενικά να έχουν μια μεγαλύτερη προστασία. Θα επαναλάβω και κάτι που σας έχω πει πολλές φορές και με αυτό θα τελειώσω. Όταν κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι την ε, Συρία, σκέφτομαι τα παιδιά, όχι τόσο τους στρατιώτες, τους μεγάλους και έχω την αίσθηση ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή με τη Γενέβα 2 στην ημερήσια διάταξη, με το COVID-2 στις 15 Ιανουαρίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα, υπάρχει μια κινητοποίηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να πιέσουμε και να δημιουργηθεί όρεξη για την ειρήνη και συγχρόνως να προσφέρουμε στήριξη στα θύματα της σύγκρουσης αυτής και ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά της Συρίας που είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ανοικοδομήσουν τη χώρα όταν σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αυτοί λοιπόν πρέπει να πάρουν βοήθεια μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και τελειώνω λέγοντας ότι ηθικά είναι ορθό να βοηθήσουμε το λαό της Συρίας. Ηθικά είναι σωστό να βοηθήσουμε το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ, ε, την Τουρκία. Αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι και προς το δικό μας το συμφέρον, γιατί αν δεν δράσουμε αποφασιστικά τώρα, τότε μια έκρηξη στην περιοχή αναπόφευκτα θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες, τραγικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κύρια για μας εδώ στην Ευρώπη. Οπότε και για ηθικούς λόγους, αλλά και γιατί είναι προς το δικό μας το συμφέρον, πρέπει να κινητοποιηθούμε και να δράσουμε. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, madame. Ευχαριστούμε πολύ κυρία πίτροπε για την τόσο ζωντανή μαρτυρία σας. Δίνω τώρα το λόγο στον ε, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπεύθυνο για τα θέματα ανθρωπιστικών ζητημάτων και θέματα έκτακτης βοήθειας την κυρία Βαλερή Άμος. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συμπρόεδρε για την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα. Όπως είπε η κυρία Επίτροπος Γεώργιεβα προηγουμένως, Πρόκειται για μια κρίση, η κρίση της Συρίας, αλλά ο ε, Συριακή κρίση αναφέρεται, αλλά είναι ουσιαστικά μια περιφερειακή κρίση με μεγάλες επιπτώσεις για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια και με σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση μέσα στη Συρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 12.200 ε, ένοπλες ομάδες που λειτουργούν, πολλές από αυτές με μαχητές που έχουν έρθει από έξω από τη Συρία, πολλοί από αυτούς τους μαχητές έρχονται και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε επίσης και τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις ροές προσφύγων από τη Συρία προς τις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος κυρία Γεώργιεβα μας έδωσε τα στοιχεία Πέραν όμως αυτών των στοιχείων θα πρέπει να κατανοήσουμε και την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων μέσα στη Συρία, οι οποίοι και αυτοί επηρεάζονται από την κρίση αυτή. Υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης και επιμελητιακές δυσκολίες για να πλησιάσουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια στη Συρία. Όλα αυτά απαιτούν καινοτόμες λύσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις κοινότητες. Είναι κάπου 250.000 άτομα σε περιοχές υποπολιορκία που δεν μπορούμε να τις φτάσουμε. Και 2,5 εκατομμύρια άτομα που είναι σε περιοχές για τις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση. Εκατομμύρια άτομα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε χώρες υποδοχής που επηρεάζονται επίσης. Σαν αποτέλεσμα χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις και αυξήσεις χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες όλων αυτών των ομάδων του πληθυσμού το 2014. Περίπου 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια που ξεπερνούν τις, τα διαθέσιμα κονδύλια και σημαίνουν έλλειψη χρημάτων για να αντιμετωπίσουμε άλλες κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα χρήματα όμως αυτά είναι απαραίτητα αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια, παιδεία, ε, υγειονομική υπερίθαλψη, υδροδότηση, και υγειονομικέ ε, ρυθμίσει για όλα αυτά τα άτομα. Εμεί έχουμε καταφέρει να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση παρά ένα αντίξω περιβάλλον ασφάλεια μέσα στη Συρία. Το πρόγραμμα διατροφή μας, παραδείγματο χάρη, έχει διαθρέψει 3,4 εκατομμύρια άτομα. Πάνω από 10 εκατομμύρια έχουν τροφοδοτηθεί με καθαρό νερό. Έχουν εμβολιαστεί. Κινητές ομάδες ιατρικού χαρακτήρα έχουν φτάσει περίπου 2 εκατομμύρια άτομα με βασικά φάρμακα. Όλα αυτά όμως δεν επαρκούν αν λάβουμε υπόψη την έκταση της κρίσης. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και την υποστήριξη συγκεκριμένα αυτού του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κέρια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας για το μέλλον. Ο λαός της Συρίας και των γειτονικών χωρών το αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον ύπατο ε, εκπρόσωπο, ύπατο αργοστή για τους πρόσφυγες, τον κύριο Αντώνη Κουτιέρης, για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από χθε είχαν καταγραφεί 2.375.000 πρόσφυγες στις γειτονικέ χώρες. Πάνω από μισή από τους πρόσφυγες αυτούς είναι παιδιά. Δεν έχω δει ποτέ παιδιά τόσο τραυματισμένα από τη βία όσο αυτά που είδα στην Συρία. Είναι περισσότερες οι γυναίκες από τους άνδρες πρόσφυγες και οι περισσότεροι άνδρες που είδα ήταν θύματα βιασμού και άλλες μορφής σεξουαλικής βίας που ήταν απόλυτα αποτροπιαστικές και απαράδεκτες. Τα άτομα αυτά χρειάζονται τρόφιμα, προστασία, στέγαση, νερό, υγειονομική περίθαλψη. Όλοι μας κινητοποιούμαστε για να τους βοηθήσουμε, αλλά υπάρχουν κενά χάσματα. Και όταν έρχεται ο σκληρός χειμώνας βλέπουμε όλα αυτά τα κενά όταν μόνο το 1 τρίτο των παιδιών βρίσκονται στο σχολείο και όταν πολλοί από αυτούς <clears throat> βασανίζονται ακόμα μετά και από την προσφυγιά από τη χώρα που έχουν φύγει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των ατόμων γιατί οι γειτονικέ χώρε δεν έχουν ανοίξει τα σύνορά του. Αλλά και με το να ανοίξουν τα σύνορά του αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν τι απαραίτητε υπηρεσίε. Βλέπετε παιδική εργασία, βλέπετε πρόορους, και πρόορους γάμους, βλέπετε πορνεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υποστηρίξει κανείς τον πληθυσμό της ε, Συρίας και της χώρες υποδοχής των προσφύγων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η επίπτωση στην οικονομία, στην, στην κοινωνία και την ασφάλεια των χωρών αυτών. Ο Λίβανος σήμερα έχει 25% του πληθυσμού του που είναι πρόσφυγες από τη Σύρια. Ήμουνα πρόσφατα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου, κοντά στην περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι μάχες στο, κοντά στο δρόμο μεταξύ Χόμς και Δαμασκού και σε ένα μικρό, σε μια μικρή πόλη ήταν πιο πολύ οι Σύριοι από τους Λιβανέζους εκεί. Όλα αυτά είναι εξολοθευτικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε χώρα. Χωρίς εξωτερική βοήθεια κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις πίεσεις. Υπάρχει και ένας ηθικός αποχρόν λόγος, όπως είπε και η κυρία Τζόζεβα αλλά είναι και θέμα δικού μας συμφέρον, συμφέροντος, γιατί η σύγκρουση περνάει όλο και περισσότερο στον ε, Λίβανο. Είναι και στο Ιράκ που έρχεται αυτή η σύγκρουση με τη σύγκρουση Ισία και Σούνη. Υπάρχει ο πληθυσμός των Παλαιστινίων προσφύγων, υπάρχουν οι χώρες του Περσικού κόλπου που επηρεάζονται και αυτές από την κρίση αυτή. Υπάρχει κίνδυνος πραγματικά ανάφλεξη στην περιοχή, όπως είπε η Επίτροπος κυρία Τζόζεβα. Έχουμε χιλιάδες μαχητές που πολλοί από αυτούς έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν γυρίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα γίνει. Και αν δεν δοθεί λοιπόν υποστήριξη στους πρόσφυγες που είναι μέσα εσωτερικά εκτοπισμένοι οι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες αν η διεθνή κοινότητα δεν κάνει κάτι για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, όλοι θα πληρώσουμε ένα πάρα πολύ υψηλό τίμημα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκουτέρες, ακολουθεί ο εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF, ο κύριος Άντωνι Λέικ. Oh, sorry. There Με συγχωρείτε. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική καταστροφή που συνεχίζει να διωγγώνεται πολύ γοργότερα από ότι εμείς είμαστε ικανοί να την αντιμετωπίσουμε. Η ανθρώπινη αυτούργοι αυτής της καταστροφής θα έπρεπε να ακούσουν κάποιους να τους λένε ότι φτάνει, φτάνει μετά από τρία χρόνια πόνου και καταστροφής Έχουμε πάνω απ' όλα μια κρίση με τα παιδιά της χώρας και ευχαριστώ Επίτροπε που το, ε, που το θίξατε. Μισό εκατομμύριο παιδιά έχουν πληγεί από την ε, κατάσταση αυτή. Ένα εκατομμύριο παιδιά είναι πρόσφυγες στις γειτονικέ χώρες με συνθήκες φτώχειας, ανισότητας και τρία εκατομμύρια παιδιά και εντός Συρίας και πρόσφυγες έξω από τα σύνορα της χώρας δεν μπορούν να πηγαίνουν συστηματικά σχόλιο. Αυτά είναι μόνο αριθμοί αλλά είναι και άνθρωποι. Το καθένα είναι ένα παιδί που θα μπορούσε να είναι ο γιο σα, η κόρη σα η το εγγονι σα. σκεφτειτε να μεγαλωνει κανεί αυτέ τι συνθήκε. σκεφτειτε η κορη σα να μην μπορεί να πάει στο σχολείο. Να μην μπορεί να μάθει και να χτίσει το μέλλον τη. Μερικά παιδιά κλαίνε από τη στιγμή που θυμούνται τις πρώτες τους εικόνες και έχουν τις πρώτες τους αναμνήσεις. Φαντάζεστε πώς είναι να μεγαλώνει κανείς έτσι. Πώς μπορούν τα παιδιά αυτά να ζήσουν στις σκηνέ στις οποίες αναγκάζονται να καταφύγουν. Ενώ υπάρχουν άθλιες συνθήκες υγιεινής και η απειλή ασθενειών που καραδοκούν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει τα παιδιά αυτά να μην ξεχνάμε ότι χρήζουν προστασία. Αυτή και η ίδια η χώρα και το μέλλον της. Το μέλλον της Συρίας θα το χτίσουν τα παιδιά της χώρας. Παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ε, παιδεία, προστασία, εμβόλια, το παιχνίδι που θε, τους αξίζει και την ευκαιρία που κάθε παιδί αξίζει να μπορεί να φτιάξει τη ζωή του. Θα καταφέρουν να μεγαλώσουν, θα φτάσουν στην ηλικία και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσει κάποια στιγμή να ξαναχτιστεί η χώρα τους όταν επιστρέψουν στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώ και η έννοια τη συμφιλίωση που θα πρέπει να έχουν στι καρδιέ του, διότι αν η απάντηση σε όλα αυτά είναι όχι, υπάρχει κίνδυνο να χαθεί αυτή η γενιά ε, των παιδιών τη Συρία ε, μέσα στην απελπισία και την ε, κατάθλιψη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι θα γίνει σε μια χώρα με παιδιά που δεν θα έχουν τι δυνατότητε που του δίνει η παιδεία και την συναισθηματική ανθεκτικότητα, πώς θα μπο... θα μπορέσουν να πετύχουν ε, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μιλάμε για θυμωμένους νέους, ε, δυστυχισμένα παιδιά που έγιναν θυμωμένοι νέοι και πιστεύουν ότι η βία είναι αναπόφευκτο κακό. Μιλάμε για εκμετάλλευση του ανθρώπου, για ένοπλες ομάδες και δίψα για εκδίκηση. Αυτό θα είναι το μέλλον της Συρίας. Χωρίς εναλλακτικές λύσεις, ο θυμός και η αγανάκτηση των μελλοντικών γενεών θα αποσταθεροποιήσουν μια ήδη ευάλωτη περιοχή και θα εξαπλωθεί η σύραξη ε, και σε άλλες περιοχές. Οι κυβερνήσεις που αποδέχονται τους πρόσφυγες, η UNICEF και οι δικοί μας φορείς φροντίζουν τα παιδιά όσο μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία με ειδικέ τάξεις, με συμβουλία από επαγγελματίες, με εμβόλια κατά της πολιομελίτιδας, με προσφορά τροφίμων και θρεπτικών συστατικών. Προσπαθούμε να σώσουμε παιδιά και ζωές, αλλά κυρίως να χτίσουμε το μέλλον της χώρας και της περιοχής. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε για μας είναι σημαντικό όχι μόνο για εκείνα τα παιδιά, αλλά για όλους μας. Για κάθε άνθρωπο στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Διότι το μέλλον αυτών των παιδιών είναι κάτι που αφορά όλους μας και έχουμε λόγο και εμείς σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο, ευχαριστώ όσους εκπροσωπούνται εδώ, ευχαριστώ για τη διαρκή σας στήριξη προς, τις, ε, προς τους φορείς του ΟΗΕ και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρούν επί τόπου και προκειμένου να πετύχουμε κάτι μαζί με τις ε, υπόλοιπες κυβερνήσεις και τη UNICEF. Ευχαριστούμε για τη στήριξη προς την οργάνωσή μας. Ευχαριστούμε για την ε, υποστήριξη των παιδιών υπέρ των οποίων όλοι εργαζόμαστε. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λέικ. Και τώρα εκτελεστική διευθύντρια του, του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος, η κυρία Κουζά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε Ζολή, Πρόεδρε Προβέρα, ευχαριστώ ε, Επίτροπε Γεωργίεβα. ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε το Σεπτέμβριο, η κρίση της πείνα, του λοιμού στη Συρία έχει επιδεινωθεί. Όταν μιλήσαμε τότε, μιλούσαμε για 3 εκατομμύρια. Τώρα θα μπορέσουμε να διαθρέψουμε 4 εκατομμύρια. Οι ανθρωπιστικέ ανάγκε και οι υπεύθυνοι για τα ανθρωπιστικά θέματα έχουν πολλέ δυσκολίε στην περιοχή. Πρέπει όμω να βρούμε νέου τρόπου για να ανταποκριθούμε στι ολοένα αυξανόμενε ανάγκε. Θα πρέπει να καταγράψουμε σωστά τις επιστηστικές ανάγκες της Συρίας και να φροντίσουμε τα αποθέματά μας. 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω έλλειψης τροφίμων και άλλου είδους βοήθειας. Για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά πρέπει να αυξήσουμε την παρουσία μας επί τόπου και να παρακολουθήσουμε το αποτύπωμα που αφήνουμε. Τον επόμενο μήνα θα εντείνουμε τις προσπαθίες μας καθώς θα φτάσουμε τα 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους ε, στη διατροφή. Αλλά επειδή υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης, ε, κάθε στιγμή που υπάρχει διανομή τροφίμων υπάρχει και κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες ε, πρόσβασης που υπάρχουν και να τις λάβουμε υπόψη μας. Λόγω χάρη, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες στη Χάσικα με την UNICEF και την έμπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, στέλνουμε τα τρόφιμα δια της ε, ε, εναέριας οδού. Είναι πολύ δύσκολο, είναι δαπανηρό το μέσο αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φτάσουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη τα τρόφιμα στην περιοχή. Όπου μπορούμε λοιπόν να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, θα το κάνουμε στη Συρία το Φεβρουάριο, ένα πρόγραμμα ε, επιστημιστικό για σχολεία θα καλύψει 350.000 παιδιά και το ίδιο για νεογνά, 15.000 εθελάζονες μητέρες και τα βρέφη τους. Στις ε, απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των προσφύγων και των κοινοτήτων ε, της χώρας που υποδέχεται τους πρόσφυγες για τα τρόφιμα, τη στέγη και την ε, υγειονομική κάλυψη. Και κάποιε φορέ είναι οι χώρε υποδοχή που αναγκάζονται να υπομισθούν αυτή την ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να καλύψουμε 2,9 εκατομμύρια πρόσφυγε, καθώ και ευάλωτε οικογένειε αυτών που υποδέχονται του πρόσφυγε. Αυτό θα είναι και η ραχοκοκαλιά τη περιφερειακή μα παρουσία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και από την άποψη του κόστου και να φροντίσουμε και τι τοπικέ οικονομίε ώστε να μην καταρρεύσουν. Είναι πολλά τα εκατομμύρια δολάρια που ε, στείλαμε στις οικονομίες της Τουρκίας, ε, του Ιράκ, της Αιγύπτου. Όλες οι προσπάθειες είναι δαπανηρές και πολύ ε, εντατικές, απαιτητικές, αλλά χάρη και στην στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάναμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε. Γι' αυτό λοιπόν να εκφράσω τις επίσημες ευχαριστίες μου προς εσάς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή της κρίσης αυτής η δική σας πολιτική βούληση και στήριξη έχει σώσει ζωές. αν θα μπορέσουμε να θρέψουμε τους πεινασμένους, τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι θύματα των αποτυχημένων πολιτικών μας λύσεων, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Το να συνεχίσουμε τη δουλειά μας είναι απαραίτητο και αυτέ οι ανάγκε θα μεγαλώνουν όσο δεν βρίσκεται πολιτική λύση. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ τη διαρκή σα βοήθεια προκειμένου να κινητοποιήσουμε νέου πόρου και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι ε, άνευ προηγουμένου ανάγκε που αντιμετωπίζουμε. Αλλά ζητούμε και την διαρκή σα υποστήριξη να κάνετε εκκλήσει κι εσεί ω προ την πρόσβαση προκειμένου να καλύψουμε τι ανάγκε όσων απελπισμένα χρειάζονται τη βοήθειά μα. Και πάνω απ' όλα θέλουμε τη διαρκή σα υποστήριξη προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πολιτική λύση. Ο Νέλσον Μαντέλα είπε ότι όλα φαίνονται αδύνατα μέχρι όμως να γίνουν. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζορτάν Ριάν έχει τώρα το λόγο που είναι διευθυντής του Γραφείου Πρόληψης Κρίσεων και του Προγράμματος των Αναπτυξιακών των Ηνωμένων Εθνών είναι επόμενο ο μιλητή μα. Σε ευχαριστώ, συμπρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω την, την ε, αναπτυξιακή διάσταση στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Τι γίνεται με την ανάπτυξη στην ε, Συρία και τις γείτονες χώρες, που βρίσκεται σε κίνδυνο βέβαια. Πάμε πίσω 35 χρόνια ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε ένδια. Τα σπίτια καταστρέφονται, οι αποταμιεύσεις χάνονται, η ανεργία έχει φτάσει στο 50% τώρα. Η χώρα έχει χάσει 2,3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Οι γείτονε χώρες με τους πρόσφυγες που υποδέχονται αλλάζουν και δημογραφικά, αλλά δημιουργούνται και κοινωνικές εντάσεις υπάρχει ανταγωνισμός για τους περιορισμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι. Η κοινωνία βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση και οι εντάσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό που χρειάζεται και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Ελπίζουμε η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και τις κυβερνήσεις να φροντίσουν για ανθρωπιστικά μέτρα επικεντρινόμενοι στην ε, προστασία προκειμένου να κρατηθεί η κατάσταση όσο γίνεται περισσότερο σε ανοιχτά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να συνεργαστούν. Η κατάσταση επίγει οι ανθρωπιστικές προσπάθειες πρέπει να γίνουν τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και μακροπρόθεσμα, αλλά ξεκινώντας βέβαια τώρα, να υπάρξει ανάπτυξη. Στην έρημο του Σαχέλ το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτό. Έπειτα πρέπει να στηρίξουμε τη δουλειά των κυβερνήσεων και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Να μην τις αντικαταστήσουμε εμείς. Πρέπει να γίνουν επίσης προσπάθειες στον κοινωνικό τομέα με προσπάθειες για κοινωνική συνοχή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ζωτική σημασία ρόλο να παίξει, συνεχίζοντας να επικεντρώνεται στη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι θα βρουν τον τρόπο να ακουστεί η φωνή τους, αλλά να είναι μια φωνή και από τους τρεις μαζί υπέρ της αναπτυξιακής προσπάθειας, ώστε η κρίση αυτή να αποτελέσει συγχρόνως και την ευκαιρία για να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται ελπίδα. Χρειάζονται μια υγιή κοινωνία, χρειάζονται ευκαιρίες, χρειάζονται προστασία και δύναμη για να αλλάξουν τις ζωές τους. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πιέρ Δημό, Γενικός Γραμματέας της Εξωτερικής Υπηρεσίας ε, τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μάλλον εξωτερική δράση. Για τρία λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να ακούμε τι έχουν να πούν οι άλλοι. Όλοι αυτοί που μίλησαν γνωρίζουν περί ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ εγώ είμαι διπλωμάτης, οπότε δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Θέλω τρία πράγματα να σημειώσω. Πρώτον, από ό,τι όλοι αντιλαμβανόμαστε εδώ σήμερα, η ανθρωπιστική κατάσταση και η ανθρωπιστική αρρωγή δυσκολεύεται όλο και περισσότερο. Κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ελέγχου. Τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα το δείχνουν. Τα είπε η Επίτροπος Γιώργεβα ότι 6,5 δισεκατομμύρια ποτέ δεν έχουμε δώσει τόσα. Συνεπώς, Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι μόνο πολιτικά μπορεί να βρεθεί μια λύση. Η λύση δηλαδή θα είναι πολιτική. Μια πολιτική λύση θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αδιανόητη κατάσταση και τόσο τραγική. Συνεπώς, τίθεται το θέμα της διάσκεψης για Νέβη 2 και κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι θέλετε να κάνω κάποιες προβλέψεις, αλλά είμαι διπλωμάτης και οι διπλωμάτες ποτέ δεν κάνουν προβλέψεις. Αλλά ας το πω ως εξή. Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας, κατά τις οποίες πρέπει όλοι όσοι θα συμμετέχουν στη Γενέβη 2 να δεσμευτούν ότι η Γενέβη 2 θα είναι επιτυχία. Αν καταφέρουμε να βάλουμε τη διαδικασία στα βλάκια, πράγμα το οποίο θα είναι δύσκολο, αλλά αν αυτοί που πάνε στη Γενέβη αρχίσουν, βοηθήσουν, αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, τότε θα έχει μπει διαδικασία στο βλάκι, πράγμα το οποίο θα αλλάξει την κατάσταση. Ήδη αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Έπειτα βέβαια, αν αυτό το καταφέρουμε και αν επιτέλους έχουμε την αρχή της διαδικασίας Γενέβη 2, τότε μπορούμε να πάμε στα διάφορα μέτρα νοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και τώρα βέβαια μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να περιμένουμε, αλλά τότε θα μπορούμε καλύτερα να πιέσουμε ε, το καθεστώς στη Συρία, την αντιπολίτευση, να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ανθρωπιστικές ε, ε, κρίσεις περί πολιτικών κρατουμένων κλπ. Μια τέτοια διαδικασία, αν μπορέσει να ξεκινήσει, αυτό θα είναι σπουδαίο. Χωρίς λοιπόν να κάνω καμία πρόβλεψη, λέω ότι έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, πολύ σημαντικό για το μέλλον της Συρίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους συνομιλητές μας για τις ε, παρεμβάσεις τους και για το γεγονός ότι μας κάνουν να κατανοήσουμε πόσο Αδύνατο είναι να δεχτούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα τώρα να ανοίξω τη συζήτηση στα μέλη των επιτροπών μας. Για δύο λεπτά ξεκινώ με την κυρία Δεκέζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που συγκεντρώσατε αυτό το τόσο ποικίλο πάνελ που μας έφερε τόσες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστώ την κυρία Γεωργία επίσης για όλες τις προσπάθειες που καταβάλει εδώ και μήνες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρώτο σημείο, όπου έχω μια ερώτηση, αφορά τον κύριο Δημό. Κύριε Δημό, μας περιγράψατε το τι γίνεται στη Γενέβη 2 και είπατε ότι είναι μια διαδικασία διέξοδη από πολιτικής άποψης. Εκεί όμως μπορεί να περιέχονται πτυχές όπως η στεγνωτική διάδρομη, η κεχηρία. Είναι μια εναλλακτική γενεβιδίο. Δεν φαντάζομαι ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ως προς αυτό. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα one shot, μια λύση δηλαδή πιο οριστική ή κάτι άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι μια πολιτική λύση για τον ε, Μπασάρ πρέπει να είναι αυτό που θα ε, κυριαρχεί στο προσκήνιο. Συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να οδεύσουμε προς μία επίλυση που να συμπεριλαμβάνει απαντήσεις, όχι αναγκαστικά αποτρεπτικές ή όλα αυτά που σχολιάσαμε εδώ, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια από τις επιλογές που έχουμε στη διαδέση μας σήμερα μπορεί να ε, προκριθεί. Διότι όταν ακούω τους ήρους προσφύγους που βρίσκονται γύρω μου, που ήδη έχουν φτάσει στο Βέλγιο, είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιφυλεκτικοί ως προς το Γενέβη 2 και το καταλαβαίνω, δεν κρίνω, καταλαβαίνω τη σημασία που έχει η συμμετοχή όλων. Αλλά εάν μιλάμε για το ανθρωπιστικό πρόβλημα είναι διαφορετικό αυτό από την πολιτική λύση. Μην πέσουμε λοιπόν σε αυτή την παγίδα. Θα πρέπει η ανθρωπιστική κατάσταση να τεθεί υποτάπητος. Είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό αυτό. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το υπόλοιπο πάνελ. Ξέρουμε ότι οι πρόσφυγες Μάλλον οι ανάγκες ξεπερνούν τον αριθμό των προσώπων που μπορούμε να καλύψουμε. Μιλήσατε κυρία Κουζάν για τα δελτία που μοιράζονται, μιλήσατε για τον ανταγωνισμό μεταξύ φτωχών οικογενειών. Ε, έχει φτάσει ο χειμώνα όταν πήγα στο Λίβανο και στη Συρία πριν από τρει μήνε. Ήδη είχαν αρχίσει να τσακώνονται μεταξύ του οι οικογένειε για το αν θα πάρουν βοήθεια ή όχι. Τελικά υπάρχει τέτοιο πρόβλημα σήμερα. Και αν ναι, Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται σωστά η κατανομή της βοήθειας. Ποιες είναι οι οικογένειες που δικαιούνται και αυτές που δεν δικαιούνται τη βοήθεια. Βάσει ποιων κριτηρίων. Πρόεδρος, ο κύριος Βέγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα, κύριε Βιλμότ, ότι είσαστε ο μόνος ομιλητής που δεν χειροκροτήθηκε. Εγώ σας χειροκροτώ, διότι μιλήσατε για ειρήνη και ειρηνικά μέσα επίλυσης της κρίσης. Σας επενώ όμως, διότι αυτό το λέτε εδώ και τρία χρόνια που διαρκεί αυτή η σύραξη, εγώ κάνω το ίδιο, αλλά είμαστε λίγοι. Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που πίστεψαν στον πόλεμο, που πίστεψαν στις φρικτές απλουστεύσεις ως προς το πρόβλημα της Συρίας και πίστεψαν ότι με μία και μόνη κίνηση μπορεί κανείς να απαλλαγεί από το καθεστώς και ότι αυτό θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα τη τόσο πολύπλοκης αυτής χώρας. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή. Και βεβαίως, προφανώς η καταστροφή αυτή απαιτεί τη μέγιστη δυνατή αφοσίωση και γενναιοδορία από πλευρά μα. Όμως αυτή είναι η συνέπεια. Είναι η συνέπεια του γεγονότος ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυτικές χώρες, όλοι από κοινού δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματική πρόκληση. Κλείνουμε τα μάτια μας, εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματική δυνατότητα. Οι Αλκάιντα και άλλοι εξτρεμιστές να αναλάβουν την εξουσία στη Συρία. Θυμάμαι κάποιος ε, μου έλεγε πριν από δύο χρόνια όταν τον έφερα ότι με κατηγόρησε ότι έχω φαντασιώσεις και οράματα. Η Αλκάιντα ποτέ δεν θα φτάσει στη Συρία. Αποκλείεται. Τώρα έγινε. Κύριε Βίλμοντ, ελπίζω ότι θα συνεχίσετε τις διαρκείς προσπάθειες υπέρ της ειρήνης και πραγματικά θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν η Ευρώπη εδώ έπαιζε έναν ε, σημαντικότερο ρόλο στην όλη ειρηνιστική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Νόησορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις ε, εκθέσεις που μας δώσανε σήμερα που άξιζε τον κόπο να, ακούσουμε. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα πιο έντονα από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Έχουμε τα έγγραφα τα οποία έχουν προέλθει από την ε, Κομισιόν και όλα αυτά δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η δέσμευση της Κομισιόν. Έχουμε και ένα κατάλογο για τα κονδύλια που δόθηκαν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Ίσως θα μπορούσαμε να συζητούμε αν κάποιο κράτος θα έπρεπε να δίνει περισσότερο ή άλλα λιγότερο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ανθρωπιστική παρέμβαση που είναι απαραίτητη. Έχουμε ένα μηχανισμό για τη διάσωση των τραπεζών. Δεν έχουμε ένα μηχανισμό όμως για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό πρέπει να είναι ένας μεσοπρόθεσμος στόχος που θα πρέπει να επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο στοιχείο, δεν έχουμε δυστυχώς κανένα κατάλογο των κρατών μελών για το πόσους πρόσφυγες έχει υποδεχθεί κάθε χώρα. Μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ε, προσφύγων που έχουν πάει στην Τουρκία, στο Ιράκ, στο Λίβανο και την Ιορδανία. Αυτό είναι όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είπε ότι θα πέρασε από 5.000 σε 10.000 ίσως περισσότερους πρόσφυγες ε, από τη Συρία. Αυτό είναι σταγόνα εν το ωκεανό όμως. Θα πρέπει όμως όταν λέμε ότι πρέπει να κατονομάσουμε και να επονιδίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και στα κάτι μέλη. Δεν χρειαζόμαστε μια δεύτερη λαπεντούσα. Πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο να γίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματική ανθρωπιστική ε, καταστροφή που απειλεί τόσο κόσμο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Συνεχίζοντας αυτά που είπε ήδη ο κύριος Νόιζα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντώνη Κουτέρες το εξής ερώτημα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στα στατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία, στα σύνορα της Συρίας. Ήδη πέρσι το Φεβρουάριο ήμασταν εκεί. Έκτοτε <clears throat> αυτός ο καταβλισμός έχει επεκταθεί σημαντικά. Ξέρω ότι μαζί με την κυρία Τζόρτζεβα ε, επισκεφτήκατε και τα, τους καταβλισμούς της, της αρμοστίας για τους πρόσφυγες στη Βουλγαρία, όπου όμως και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αποτροπιαστική. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του κύριου χρηματοδότε τη υπάτη αρμοστία για του πρόσφυγε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορείτε όμω να μα πείτε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, πού βρίσκονται οι ευθύνε μα, με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε του Ιορδανού, του Τούρκου, του Λιβανού, τους Ιρακινούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά στέγασης και διατροφής όλων αυτών των προσφύγων από τη Συρία και τι ακριβώς περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γουτέρες όταν πρόκειται για τη βοήθεια για το πρόβλημα της κρίσης των Συρίων προσφύγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Γκουτιέρες, η ανθρωπιστική κρίση δεν θα λήξει ποτέ αν δεν λήξει ο πόλεμος. Οπότε ρωτάω τον κύριο Γκουτιέρες αλλά και όλους εσάς που έχετε βρεθεί εκεί. Τι μαθήματα παίρνει κανείς τι μπορείτε να μας μεταφέρετε από εκεί ώστε να βρούμε μια πολιτική λύση, ώστε η Γενέβη 2 να προχωρήσει και να συμμετέχουν εκεί όλες οι πλευρές. Η συμφωνία, για παράδειγμα, με το Ιράν είναι κάτι που μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις ώστε να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι διάφορες πλευρές στη Γενέβη. Φυσικά καταλαβαίνω ότι χρειάζεστε χρήματα για να αντιμετωπιστεί η τραγική κατάσταση της κρίσης, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να βρεθεί η πολιτική λύση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Φένσον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχουμε εδώ ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται γνωρίζουν από πρώτο χέρι την κατάσταση. Κάποιος είπε ότι αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή. Μα είμαστε μέσα στην καταστροφή. Υπάρχουν ακραίες ομάδες που συμμετέχουν ε, εκεί στη σύγκρουση με μεγάλη βία. Έχουμε την εντύπωση νομίζω ότι 22 Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία η σημαντική. Αλλά ας σκεφτούμε τι θα γίνει μετά στις 22 Ιανουαρίου επίσης. Μιλώντας δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές φανατικές ομάδες και θα ήταν σωστό να πούμε ότι αυτούς δεν τους νοιάζει το τι θα αποφασίσουμε εμείς στη Γενέβη. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι φανατικές ομάδες θα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί επί τόπου, ό,τι και αν αποφασίσουμε εμείς στις 22 Ιανουαρίου. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ απεσιόδοξα, κύριε Πρόεδρε, αλλά πώς μπορεί κανείς να μην είναι απεσιόδοξος έτσι όπως έχει κατάσταση σήμερα. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρο. Η κυρία Λιπτσεβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ που την οργανώσατε. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα για να συζητήσουμε. Για τους πρόσφυγες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλα πράγματα. Εδώ δεν τα λέω αυτά προσωπικά για κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα σκεφτούμε. Πώς να διακρίνουμε το θέμα των προσφύγων από τους παράνομους μετανάστες, γιατί είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα. Επίτα, πώς να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες, τις γείτονες χώρες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό των προσφύγων. Επίσης, πολύ θα θέλαμε συγκεκριμένες προτάσεις από εσά. Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε βέβαια για την ειρήνη, για τις αρχές, ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, αλλά θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Κουτιέρες, εσείς έχετε έρθει στη Βουλγαρία, ξέρετε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Ίσως το ίδιο να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Θα είχατε να σχολιάσετε κάτι και έχετε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα σε χώρες όπως είναι η δικιά μου. Γιατί είναι μια χώρα που περάζεται πολύ από αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κύριε Λάτφορτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έρχεται μετά από την ερώτηση της κυρίας Ατζεντίνη και μάλλον απευθύνεται στον κύριο Γκουτιέρες πιο πολύ. Να ρωτήσω περισσότερες λεπτομέρειες μετά από αυτό που ρώτησε και εκείνη, δηλαδή τι έχει να συμβουλέψει τις χώρες μέλη ο κύριο Γκουτιέρε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κρίση με το θέμα των προσφύγων συγκεκριμένα. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες των χωρών που προσπαθούν να υποδεχτούν πρόσφυγες, είτε δίνοντας ανθρωπιστική βοήθεια, είτε σε καταβλισμούς, η άποψή σας ποια είναι, τι νομίζετε ότι μπορεί να προσφέρει η κάθε χώρα, πώς μπορεί να βοηθήσει στο θέμα των προσφύγων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Γενικός μας Διευθυντής, ο κύριος Στέφανο Μασεβίση, που είναι Γενικός Διευθυντής της HOME για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή που μου δίνετε. Η Επίτροπος Μάλστρομ έχει δεσμευτεί να βοηθήσει από πλευράς Υπουργών Εσωτερικών. Να συμπληρώσω και εγώ λίγο τα νούμερα. Σήμερα έχουμε 65.000 Σύριους οι οποίοι έχουν το καθεστώς πρόσφυγα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011 δηλαδή όταν ξέσπασε η κρίση και βρίσκονται κύρια σε δύο χώρες μέλη, στη Γερμανία και τη Σουηδία και σε άλλες χώρες αλλά κυρίως η μεγάλη συγκέντρωση είναι εκεί. Και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία σε αυτές τις δύο χώρες θέλουν να πάνε. Έρχονται, φτάνουν και αεροπορικά και οδικός αλλά και μέσω θαλάσσης. Ξέρετε με την τραγωδία της ε, Αμπεντούσα είχαμε εκεί αρκετούς Σύριους επίσης. Γι' αυτό και βλέπουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια και της Task Force για την Μεσόγειο που έχει ήδη εκμονήσει μια πρώτη έκθεση που ελπίζω αύριο να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει απαιτούμενη υποστήριξη οικονομική δηλαδή από τις χώρες μέλη και ό,τι άλλα μέσα μπορούν τα κράτη-μέλη να προσφέρουν. Και είναι και το θέμα των καταβλισμών βέβαια, αλλά θα έρθω αργότερα σε αυτό. Τώρα ο δικός, έρχονται όλο και περισσότεροι τον τελευταίο καιρό, είναι χειμώνα, πάνε στην Τουρκία και επηρεάζουν βέβαια τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα. Σίγουρα και η Βουλγαρία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την είσοδο προσφύγων. Δεν λέμε ότι η Βουλγαρία τους ε, ζητάει να επιστρέψουν. Όχι. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες αυτούς. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τις υπηρεσίες μας, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, προσπαθούμε να βρούμε λύση. Κινητοποιούμε και πόρους. Ποτέ δεν φτάνουν βέβαια αλλά αν μη τι άλλο προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί. Το επόμενο βήμα θα είναι να αυξήσουμε την ε, απάντησή μας όσον αφορά τις 30.000 που θα χρειαστούν από ό,τι φαίνεται για τον επόμενο καταβλισμό. Στις, ε, το πρώτο εξάμεινο του 2014 θέλουμε να φροντίσουμε όχι μόνοι μας, αλλά σε συνεργασία και μάλλον δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να φανούμε στη διάσκεψη, να φροντίσουμε σε συνεργασία να βρούμε μια λύση και σε αυτό. Πάντως για τους καταβλισμούς δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης προς την Συρία, η βοήθεια που δίνουμε στη, στο Λίβανο και σε άλλες γείτονες χώρες. Μερικές φορές μια χώρα μπορεί να βοηθήσει μια άλλη που έχει πρόβλημα. οι χώρες οι οποίες αντικειμενικά βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση όπως η Βουλγαρία για παράδειγμα πρέπει να βοηθηθούν. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε και την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. 100% το λέμε ότι δεν στέλνουμε πίσω κανένα Σύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μάργκοτ Έλλης έχει τώρα το λόγο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 οι κίνδυνοι για την ασφάλειά τους στη Συρία, μαζί με το γεγονός ότι δεν έχουν δυνατότητες φύγης, έχουν φέρει τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θεωρείται τώρα ότι κάπου 270.000 Παλαιστίνοι πρόσφυγες από τη Συρία, δηλαδή το μισό τους, έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. Αυτό συμπεριλαμβάνει 140.000 πρόσφυγες οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από τις εστίες τους πριν από ένα χρόνο που ήταν κέντρο μαχών στις Συρίες. Έχουν πάει σε άλλες χώρες όπως είναι σε άλλες χώρες όπως η Ορδανία, ο, ο Λίβανος, ακόμα και στη Λωρίδα της Γάζας. Επειδή δεν έχουν νομικό καθεστώς, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν ακόμα και στα γειτονικά κράτη. Πολλοί τελικά βλέποντας ότι δεν έχουν κανένα ασφαλές καταφύγιο επιστρέφουν στη Συρία η κρίση στη Συρία έχει φέρει τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε μία ακόμα σύγκρουση όπου απλώς επαυξάνεται τα βάσανα που έχουν περάσει μετά από την αραβο σύγκρουση. Μετά από αυτές τις πολλαπλές μετακινήσεις, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες της Συρίας ψάχνουν απεγνωσμένα για να βρουν ασφάλεια σε μια περιοχή που έχει καταστραφεί από την Συριακή κρίση. Θέλω να επενέσω την κυβέρνηση του Λιβάνου γιατί έχει κρατήσει ανοιχτά τα σύνορα για τους Παλαιστίνιους ε, πρόσφυγες από τη Συρία που είναι τώρα 51.000 στο Λίβανο. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες προκλήσεις που αντιμετωπίσει αυτή η κοινότητα όταν προσπαθούν να πάνε στο Λίβανο. Έχει η επίση ζητήσει από την κυβέρνηση της Ιορδανίας να εφαρμόσει αρχές της μη επαναπρόθεσης και ίσης μεταχείρισης όλων των προσφύγων. Βρισκόμαστε στο προσκήνιο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Θέλουμε να τονίσουμε όμως την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα αυτών των προσφύγων. Εφέτος η Ούλα άνοιξε νέα γραφεία για μικροκονδύλια στην ε, Λατούς, στη Λατάκια και σε άλλα μέρη και ιδίως και στην περιοχή που έχει περισσότερο κουρδικό πληθυσμό στη Συρία. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η σταθερότητα των κοινοτήτων εκεί και να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει την εφαρμογή ανθρωπιστικών δράσεων ω τμήμα τη προορατική μα στρατηγική. Το προσωπικό μα στη Συρία εξακολουθεί να δίνει παιδεία και υγειονομική περίθαλψη μαζί με την ανθρωποστική παρέμβαση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποτροπεί ο κίνδυνος της έκθεσης στην Δία. Δυστυχώς στις 2 Δεκεμβρίου χάσαμε το δέκατο από τα μέλη του προσωπικού μας που χάνει τη ζωή του και άλλα 20 αγνοούνται. Η κατάσταση ασφαλείας εξακολουθεί να επιδεινώνεται και η ούρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να υπάρξει μια διαχείριση της κρίσης που θα υποστηρίξει τις δράσεις μας. Το 2014 έχουμε κάνει μια περιφερειακή έκκληση για 400.000 αμερικανικά δολάρια για να μπορέσει να δοθεί βοήθεια σε ευάλωτους Παλαιστίνιους προσφύγες και ζητούμε επίσης να γίνουν αυτές οι προσπάθειες με μικροχρηματοδότηση, τεχνική κατάρτιση και άλλες δραστηριότητε να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους. Για τα προγράμματα επισκεπτισμού στο σχολείο και αυτά θα προσπαθήσουν να καλύψουν τι ανάγκε τη έλλειψη διατροφή. Το Οι κοινωνικέ συνθήκε και η διαρκή επαγρύπνηση πρέπει να είναι από τι βασικέ μα παρεμβάσει ε, μαζί με τι ε, γενναίες που γίνονται. Η μάστιγα των, ε, μάλλον το βάρο των ε, σύρων προσφύγων είναι κάτι που ε, απαιτεί την προσοχή μα, Διότι το καθεστώ των σύρων προσφύγων αφορά όλου μα, αλλά και οι συνθήκε διαβίωση του. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτε ομάδε δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολο, δεν έχουν αντοχή και ανθεκτικότητα και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν στην αρχική τους, στον, αρχική τους, στον αρχικό τους τόπο προέλευσης, τους Παλαιστίνους λοιπόν πρόσφυγες πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προστασία και αφού ε, επιληθεί η κρίση της Συρίας θα πρέπει να βρεθεί παράλληλα και μια λύση για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία μου. Θα δώσω και πάλι το λόγο για τρία λεπτά στον καθέναν από τους προσκεκλημένους μας για να προσπαθήσει να απαντήσει στα μέλη του Κοινοβουλίου. Κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχολεία σας. Η ανθρωπιστική κρίση είναι το θέμα που οι περισσότεροι σχολιάσατε και ε, νομίζω όλοι επικεντρωθήκατε σε αυτό. Θα μιλήσω και εγώ λοιπόν για τρία βασικά θέματα. Κύριε Γκόμες, είπατε τι απαιτείται για να πετύχει η Γενέβη 2 και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε από την πλευρά της ανθρωπιστικής κοινότητας για να διευκολύνουμε τη λύση. δουλειά μας είναι να βρούμε το πλαίσιο το πλαίσιο, αλλά με κάποια διορατικότητα, προσπαθώντας να διαδούμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει ειρήνη. Το κάνουμε αυτό χρονιά μετά τη χρονιά. Πέρσι είπαμε ότι αν δεν υπάρξει ειρήνευση, θα αυξηθεί ο εξτρεμισμός εντός της Συρίας και περισσότεροι πρόσφυγες θα αρχίσουν να τραπετεύουν. Θα έρχονται πρόσφυγες στην Ευρώπη. Έγιναν αυτά. Επαληθεύτηκαν. Τώρα βλέπουμε πάλι την απουσία ειρήνη στο άμεσο μέλλον και καταλαβαίνουμε ότι είτε βαθμιδιαία θα επιδεινωθούν οι συνθήκε, είτε ενδεχομένω θα υπάρξει έκρηξη. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια, ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, να έχουμε ένα πλαίσιο διορατικότητας για να δούμε τι συμβαίνει στο μέλλον. Οι ανάγκες όμως πολλαπλασιάζονται και διωγγώνονται γοργότερα από ό,τι μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε. Και διαρκώς είμαστε σε καθυστέρηση βλέπουμε ότι απαιτείται πολιτική πυγμή για να βρεθούν λύσεις όπως στην περίπτωση των χημικών όπλων. Υπήρξε γενικώ ένα κλίμα φόβου με τα χημικά όπλα και εκεί αναλάβαμε δράση. Όμως οι 25.000 Σύριοι που χάσαν τη ζωή τους δεν πέθαναν ω επιτοπλίστων από τα χημικά όπλα, αλλά από συμβατικά. Ε, ε, αυτό σημαίνει ότι κάπως δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό εντό του οποίου αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι κίνδυνος μόνο για του Σύρου, αλλά για όλου μα. Σκοπό τη σημερινή συνάντηση είναι ακριβώ να ε, επιστήσουμε την προσοχή όλων σε αυτό και να αξιοποιήσουμε το τις ιδιαίτερες γνώσεις, τα φώτα του, είπα, του προσώπου Γκουτέρες, για να δούμε τι πρέπει να κάνει η ανθρωπιστική κοινότητα στο μέλλον. Ποια είναι η μελλοντική πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε δηλαδή. Δεν έχω χρόνο ήδη. Πω από 26 δευτερόλεπτα. Δεύτερον, Είπατε για τον, ανθρωπιστικό για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανθρωπιστική Βοήθεια. Στην Ευρώπη έχουμε αναλάβει μια πολύ σοβαρή δέσμευση. Όσα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσα κάνουν τα κράτη-μέλη, να τα συνενώσουμε με έναν τρόπο συνεκτικό. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα ετοιμασμένοι για να συμπληρώσουμε μεν τι προσπάθειε των ΔΕ. Αλλά οι ανάγκε έχουν φτάσει εκεί και η δική μας πόρη είναι ακόμη πιο χαμηλά. Το τι θα γίνει λοιπόν σήμερα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμά. Εμεί ενοποιήσαμε τι προσπάθειε στο ανθρωπιστικό επίπεδο και την ανάπτυξη με του ανθρωπιστικού πόρου του συνδυάσαμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι πώ οι άλλοι θα, θα εντείνουν τι δικέ του προσπάθειε. Ενώ τι χώρε του κόλπου, του Ρώσου και του υπόλοιπου. Πώ αυτοί να κάνουν πιο εντατικέ προσπάθειε χωρίς να φαίνεται ότι εμείς από τη Δύση τους κάνουμε μάθημα και τους δείχνουμε τι πρέπει να κάνουν ε, επιτακτικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει συνοχή στις προσπάθειες και όλοι πρέπει να εργαστούμε σκληρά ε, για αυτό το σκοπό. Τελευταία μου παρατήρηση, το ερώτημα που τέθηκε για συγκεκριμένες συστάσεις. Κοιτάξτε, ξέρουμε τι επιτυγχάνει. Έχουμε εδώ τον υπατεκπρόσωπο Γκουτέρες, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι. Ξέρουμε τι πετυχαίνει και τι όχι. Και είναι χαρά μας και να το μοιραζόμαστε. Στην έκκληση υπάρχουν λεπτομέρειες επιλεπτομεριών για δράσεις που προτείνονται βάσει των καλών αποτελεσμάτων που έχουν δώσει. Κατά πολέμηση της καταστροφής, ε, της ε, εκδίωξης ε, προσφύγων ναι, αυτέ τι ειδικέ γνώσει μπορούμε να τι αντιμετωπι... αξιοποιήσουμε και για τι δικέ μα τι χώρε που αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα. Και είμαι στη διάθεσή σα, αν το χρειαστείτε, να σα το προσφέρω αυτό ω γνώση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Έμο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. να κάνω μια γενική παρατήρηση καταρχήν, να μου επιτρέπετε. Πέρσι το Μάρτιο ήταν ένα εκατομμύριο άτομα στη Συρία που επλήττονται από την κρίση αυτή. Σήμερα είναι 9,2. Έχουμε μια εκθετική αύξηση των θυμάτων της κρίσης αυτής. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα παραγνωρίσουμε όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να εξευρεθεί μια πολιτική λύση. Ακόμα και αν σταματούσε αύριο ο πόλεμος στη Συρία. Ο αντίκτυπος στη Συρία και τις γειτονικέ χώρες θα χρειαζόταν χρόνια για να μπορέσει να σβήσει. Η, Συρία, η, οικονομία της ε, Συρίας έχει καταρρεύσει, το νόμισμα έχει χάσει την αξία τα σχολεία, τα νοσοκομεία έχουν καταστραφεί, κύριες υποδομές έχουν ε, καταστραφεί επίσης και τα άτομα τα οποία φύγανε, ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η διάσκεψη Γενέβη 2 θα μπορέσει να επιτύχει. Υπήρχε ένα ερώτημα για το τι έχουμε μάθει από τις επιτόπιες μας προσπάθειες για να μπορέσει να βρεθεί μια πολιτική λύση. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι απόλυτα κατεπήγον να θυμηθούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος όλων αυτών των γεγονότων στους απλούς ανθρώπους σε ό,τι αφορά την προστασία των αμάχων καταρχή, αλλά και γενικότερα. Πρέπει να θέσουμε τους ανθρώπους στο κέντρο της απάντησής μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα επιρροής που έχουμε, είτε προς την κυβέρνηση είτε προς τις αντιπολευόμενες φατρίες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή κατανόηση της ανθρωπιστικής επίπτωσης αυτών των, ε, αυτής της σύγκρουσης, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ανθρωπιστικά θέματα ως ένα δυνητικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνη μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους το πόσο μακροχρόνιες θα είναι επιπτώσεις, όσο χρονίζει αυτή η σύγκρουση, όλο περισσότερο οι ακραίες ομάδες, οι εξτρεμιστικές ομάδες θα έχουν μεγαλύτερη βάση στη χώρα αυτή και θα κάνουν πολύ πιο δύσκολη την επιτεύξη ειρήνης στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Αντώνη Κουτέρες έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και πάλι που βρίσκομαι στην κοινοβουλευτική ζωή μετά από 25 χρόνια. Υπήρχαν πολλά ερωτήματα τα οποία μου τέθηκαν. Ζητώ λοιπόν κάποια ανοχή σε σχέση με το χρόνο. Καταρχήν, το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όταν υπάρχουν περισσότερες ανάγκες από ότι πόροι. Αναφέρθηκε το θέμα της διανομής τροφίμων στο Λίβανο σχετικά. Έχουμε οργανώσει το πρόγραμμά μας μαζί με τους άλλους φορείς που δίνουν ανακουφιστική βοήθεια βάσει τριών κατευθύνσεων για να αντιμετωπίσουμε το κενό που υπάρχει. Γιατί υπάρχει κενό, δεν έχουμε αρκετή αρκετούς πόρους. Καταρχήν, να δώσουμε πρώτη προτεραιότητα στι δραστηριότητε που σώζουν ανθρώπινε ζωέ. Δεύτερον, η βελτίωση τη αποδοτικότητα. Περισσότερο χρήματα και κουπόνια από τη ηλική βοήθεια γιατί είναι πιο αποτελεσματικό. Και τρίτον, η στοχοθέτηση. Αυτό βασίζεται σε μια πλήρη αξιολόγηση η οποία είναι απαραίτητη να γίνει. <clears throat> Έχουμε εξετάσει τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού και κάνουμε κάποιες επιλογές επί τη βάση του τροτού αυτών των ομάδων. Στο Λίβανο προσπαθούμε να φτάσουμε 75% του πληθυσμού εκεί πέρα που χρειάζεται βοήθεια και στην Ιορδανία υποστηρίζουμε 35.000 οικογένειες. Αυτό είναι το μάξιμο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι δραματικό αυτό, αλλά ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες είναι να έχουμε και τα χρήματα για όλους. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τι τοπικέ κοινότητε στι διάφορε χώρε πρώτα με οικονομικά μέσα και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ενθεκτικότητα τη Ιορδανία, το Πρόγραμμα Σταθεροποίηση στο Λίβανο τα καταπιστεύματα τα οποία έχει δημιουργήσει η Παγκόσμια Τράπεζα στο Λίβανο, <clears throat> αλλά εξίσου σημαντική είναι, χρηματο... όπως και η χρηματοδοτική υποστήριξη, είναι η κατανομή του βάρους. Αυτό έχει μια συμβολική σημασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επανεγκατάσταση αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν τα άτομα αυτά να έχουν ένα μόνιμο καθεστώς προσφύγων, ανθρωπιστική αναγνώριση, με προσωρινό καθεστώς ε, προσφύγων με δικαίωμα διαμονής και εργασίες. Έχουμε ζητήσει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, έχουμε και μάλλον θέσεις ε, προσφύγων. Μέχρι 10.000 μας έχουν δοθεί από τη Γερμανία και έχουμε την ελπίδα θα αυξηθεί ο αριθμό των προσφύγων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε τα σύνορα ανοιχτά. Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα σύνορα της ε, Τουρκίας και της Ιορδανίας και του Λιβάνου και μετά να κλειστά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θέλει κάποιος να πάει κάπου αλλού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει το άνοιγμα των σύνορων. Είναι πραγματικά κάτι πραγματικά λανθασμένο όταν ένας ε, Σύρος για να έρθει στην Ευρώπη πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του σε κάποιο καραβί που διασχίζει τη Μεσόγειο. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές που θέλουμε, με την επανένωση των οικογενειών, με πάρα πολλά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν για να μπορέσουμε να δώσουν δυνατότητα σε αυτούς που χρειάζονται προστασία να έρθουν στην Ευρώπη. Πώς τους διακρίνουμε από τους παράνομους ε, μετανάστες. Μα υπάρχει μια οδηγία για, την, ε, για τις προϋποθέσεις που μας, οδηγεί, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν έχετε μια οικογένεια από τη Συρία, στα σύνορά μας υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι χρειάζονται προστασία. Δεν νομίζω ότι απλώς είναι σε αλίευση καλύτερες θέσεις εργασίας σε μια άλλη χώρα. Νομίζω ότι το βάρος της αμφιβολία, η αμφιβολία θα πρέπει να είναι υπέρ αυτών οι οποίοι ζητούν βοήθεια και άσυλο. Εναπόκειται βέβαια σε κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει πότε δίνει το καθεστώ του ασύλου και του πρόσφυγα και όχι να προστατεύσει αυτού που δεν θέλει. Η κατάσταση συγκεκριμένα στη Βουλγαρία. Τι χρειάζεται στην περίπτωση αυτή. Χρειάζεται μεγαλύτερη διεθνή αλληλεγγύη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλληλεγγύη. Ξέρω ότι έχουν δοθεί κονδύλια. Η υπάτη αρμοστία γίνεται πιο λειτουργική στην ε, Βουλγαρία δίνουμε, δίνουμε και βοήθεια, κάτι το οποίο δεν φανταζόμαστε ότι ποτέ θα πρέπει να το κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξουμε τη δέσμευσή μας και οι βουλγαρικές αρχές που είχαν την ευκαιρία να πάω μαζί με την Επίτροπο Γιώργεβα πρέπει να επενδύσουν σε υποδομές ε, εγκατάσταση των προσφύγων και στην ολοκλήρωση, στην ενσωμάτωσή τους μέσα στη βουλγαρική κοινωνία. Δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχτούν αυτό το ρεύμα προσφύγων, αλλά αυτή τη στιγμή έρχονται αυτοί οι πρόσφυγες. Αυτό όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι σαν βουλγαρικό πρόβλημα, αλλά σαν ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται από την Τουρκία ή από τη Μεσόγειο και μετά θα πάνε κατευθείαν στις χώρες της Μεσογείου που είναι πιο κοντά και οι χώρες που έχουν ε, δεχθεί πιο πολλούς πρόσφυγες από τη Συρία αυτή τη στιγμή είναι η Σουηδία και η Γερμανία και θέλω να εκφράσω την ευρωμοσύνη μου προς τις χώρες αυτές. Και για να έρθω στο ερώτημα της Άννα για μια εξέβεση πολιτικής λύσης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει και στρατιωτική λύση η οποία μπορεί να επιτευχθεί στη Συρία. Αυτό που δεν είναι σαφές για μένα είναι το κατά πόσο αυτοί που πολεμούν και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τους αντιμαχόμενους, οι λεγόμενοι εμπλακόμενοι, έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση. Ελπίζω ότι η Γενέβη 2 θα μπορέσει να πείσει και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και ελπίζω ότι γίνεται η διάσκεψη της Γενέβης 2 σε μια χρονική στιγμή που όλοι καταλαβαίνουν κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και δεν μπορεί να υπάρξει καμία πολιτική λύση αν δεν καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί κανείς να κερδίσει τη μάχη στη Συρία και ελπίζω να γίνει αυτό πολύ γρήγορα γιατί αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση όχι μόνο για την περιοχή αυτή συγκεκριμένη αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ λέει πρόεδρος. Η κυρία Πατερά Ευχαριστώ. ως εκπρόσωπος αναφέρεται στο θέμα του πώς στοχεύουμε την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά τα κριτήρια που έχουμε συμπεριλαμβάνουν ε, το μέγεθος του νοικοκυριού, κατά πόσο επικεφαλής είναι γυναίκα ή όχι, αν έχουν γη στην ιδιοκτησία τους ή αν η γη που έχουν είναι μικρής ε, αξίας ή αν υπάρχουν ανάπηρα άτομα στο νοικοκυριό. Μέσα στη Συρία υπάρχουν 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται αρρωγή και είπαμε ότι προσφέρουμε 6,5 εκατομμύρια πρόκειται κυρίως για αυτούς οι οποίοι μετατοπίζονται μέσα στη χωρα πεντε 5-7 φορές αυτοί χρειάζονται πάνω απ' όλα τη βοήθειά μας και κυρίως είναι ε, γυναίκες επικεφαλής των οικοκυριών. Η δυσκολία είναι μεγάλη γιατί μας απασχολεί και το θέμα της ποιότητας, όχι μόνο της ποσότητας. Γι' αυτό είναι δύσκολο να βρούμε σε ποιον πρέπει να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια κατά προτεραιότητα. Δεν πρέπει να νιώθουν και ότι τους αρνούμαστε τη βοήθεια. αν κάποιος νιώθει ότι έχει ανάγκη για βοήθεια, αλλά εμεί δεν το θεωρούμε τόσο ευάλωτο, παρόλα αυτά προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε και να τον προσεγγίσουμε. Τι μαθήματα παίρνουμε και μπορούν να βοηθήσουν για πολιτική λύση. Τα πανικοί συνάδελφοι. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω διαπιστώσαμε ότι το βασικό είναι να υποστηρίζουμε τον κόσμο. Όταν ε, υπήρχε το θέμα τα χημικά όπλα και η κοινωνία ζητούσε μια απάντηση στο θέμα αυτό των χημικών όπλων, βρέθηκε η λύση. Τώρα λοιπόν θα βρεθεί πολιτική λύση άμα ο κόσμος τη ζητάει. Και όταν λέω κόσμος δεν εννοώ μόνο εσάς που βρίσκεστε εδώ, εννοείται ότι εσείς πρέπει να το κάνετε και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ολόκληρη η διεθνή κοινότητα, γιατί υπάρχουν Κατάρ, Σιδική και άλλες χώρες που μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ για την πολιτική λύση, όσο και οι δυτικέ κυβερνήσεις. Συνεπώς, όλη η διεθνή κοινότητα πρέπει να ψώσει τη φωνή της και να ζητήσει πολιτική λύση και έτσι και εμείς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τζόρνταν Ριάν. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Τα καλά που συμβαίνουν σε αυτήν την μεγάλη τραγωδία είναι ότι οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται επί τόπου και δουλεύουν ηρωικά αλλά και συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους από ό,τι ποτέ η αναπτυξιακή υπηρεσία, η ανθρωπιστική, προσπαθούν να λύσουν τις ελλείψεις στον ανθρωπιστικό και τον αναπτυξιακό τρομέα. Με τις υπηρεσίες των ΗΕ λοιπόν δίνονται τρόφιμα, φτιάχνουν κουζίνες, οι άνθρωποι εκεί πρέπει να τις λειτουργήσουν αυτές τις κουζίνες. Η πατία για τους πρόσφυγες κινητοποιεί τοπικές ομάδες, ανθρώπους δηλαδή επιτόπου και διώχνουν τους ε, επαναστάτες και επιστρέφουν τον κόσμο στα σπίτια του. Οι άνθρωποι αντιστέκονται, οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τη ζωή τους πίσω στα χέρια τους, θέλουν τα παιδιά τους, ακόμα και αυτοί που καταστράφηκαν πλήρως θέλουν τα παιδιά τους να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η πολιτική λύση λοιπόν έρχεται όταν οι άνθρωποι λένε όπως είπε και τον Ηλέκ φτάνει πια, δεν θέλουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να ακουστεί φωνή τους. Και οι κοινοβουλευτικοί πρέπει να ακούσουν αυτή τη φωνή, να την ε, δυναμώσουν και να την κάνουν ακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες παντού στον κόσμο να δυναμώσουν τη φωνή αυτή και να την κάνουν ακουστεί και στη Γενέβη 2, αλλά κυρίως να υπάρξει ένα ακούραστο κίνημα σε όλο τον κόσμο που να λέει ότι η κατάσταση αυτή στη Συρία πρέπει να σταματήσει γιατί έχει κάνει τόσο κακό και γιατί θα συνεχίσει να προκαλεί καταστροφές και από περιφερειακή καταστροφή θα γίνει γενική καταστροφή. Λοιπόν υπάρχουν θετικά, επειδή όπως είπαμε οι άνθρωποι εκεί κάνουν τεράστιες προσπάθειες, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά, συνεργασία για να μπορέσει η ζωή των ανθρώπων εκεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέψατε να πάρουμε το λόγο εδώ και να ξέρετε ότι ευχαριστούμε πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να βρει πώς τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων, τα δολάρια είπε ο, ο να ξέρουμε ότι είναι μεγαλύτερη συνεισφορά ποτέ που δόθηκε σε τρεις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και που πάνε κατευθείαν για να βοηθηθούν παιδιά με τρόφιμα και πάνε και για βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Είναι συμβολικό ότι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο και το είδαμε είτε πρόκειται για το Σαχέλ είτε πρόκειται για αλλού στον κόσμο. Και θέλω να τονίσω ότι η ΕΚΟ και η Επίτροπος Γεωργεύα να ξέρετε ότι από τη θέση που είσαστε μπορείτε να προσφέρετε πολλά ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά, αλλά συγχρόνως αλλάζεται τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πραγματικότητα η αναπτυξιακή δράση. Γιατί υπάρχει συνεργασία και ελπίζουμε ότι με τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, με συνεργασία μεταξύ μας θα μπορέσουμε το 2014 και μετά να βρούμε τη λύση και να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Καλές γιορτές σε όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δημό και θα ήθελα να μας εξηγήσει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια θα μπορούσε να ασκήσει την επιρροή της σε αυτήν την σύραξη, να της δώσει ένα τέρμα και επιτέλους να βοηθήσουμε στην πολιτική και ανθρωπιστική επίλυση. Αυτό επιδιώκουμε σε καθημερινό επίπεδο κυρία Πρόεδρε. Ευθύς εξ αρχής είμαστε εκείνοι που υποστηρίζουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος ε, Ανκιμούν, ε, ο κύριος Κοφιανάν, ο κύριος Ιμπραήμι προσπαθούν να προσπάθησαν με τη σειρά τους να ασκήσουν την απαραίτητη επιρροή. Μάλιστα το 2012 δεν πάψαμε να επαναλαμβάνουμε ότι μόνο η πολιτική λύση θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος από την κατάσταση αυτή. Είχαμε διαρκείς επαφές, διατηρήσαμε την επαφή μας με τους μεν και τους δε, θα το εξακολουθήσουμε. Απλώς έχουμε την αίσθηση ότι σήμερα η πραγματικότητα αυτή, η πραγματικότητα που ισχύει στην πράξη, επιβάλλεται σε όλους. Για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Δεκεζέρ. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά όλες οι θέσεις είναι σεβαστές. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε για την ε, συνδιάσκεψη της Γενέβης και ότι ο μόνος μας στόχος δεν θα πρέπει να είναι ο κύριος Μπασάρα Λασάντ. Βέβαια το στόχο αυτό τον συμμερίζονται πολύ όμως το ερώτημα είναι πώς θα καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και όλο το ζήτημα είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα επιτρέψει ε, να περάσουμε στην μετάφαση την οποία τόσο πολύ επιθυμούμε. Να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα εμπιστοσύνης, τα οποία τα συζητήσαμε πάλι σήμερα και μέσω της συνδιάσκεψης της Γενέβης που θα μπορούσε να είναι μια ε, συνδιάσκεψη που να καλύψει και άλλα θέματα, θέματα που αφορούν διαφορετικές πτυχές του όλου ζητήματος που έχει δημιουργηθεί, όλο αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εδώ να αναφέρω την πολύ δίκαιη απορία του κ. Κουτέρες που λέει έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα θετική λύση. Έχετε δίκιο. Ε, πήρε πάρα πολύ καιρό και υπήρξε πάρα πολύ denial, πάρα πολύ άρνηση από την πλευρά πολλών μέχρι να το αντιληφθούν. Εμένα αυτό όμω που με αφορά περισσότερο σε αυτή την δραματική κρίση τη Συρίας και μα ε, πλήττει όλου στην πραγματικότητα είναι ότι όπως αλλάζουν οι ανάγκες, αλλάζουν και οι τοποθετήσεις και οι διαθέσεις των μάρκετων. Ακούω σήμερα ότι άρχισαν οι επαφές μεταξύ του Άρμη, του ελεύθερου σειρακού ε, στρατού και του επίσημου καθεστώτος της Δαμασκού. Εδώ μας λένε δυτικοί εταίροι μας ότι έχουν αρχίσει επαφές με ισλαμιστικές ομάδες. Καταλαβαίνουν όλοι τα πράγματα είναι ρευστά, εξελίσσονται, δεν παραμένουν ε, αμετακίνητα. Εάν λοιπόν πετύχει η συνδιάσκεψη Γενέβη 2, θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και την πραγματικότητα όσο έχει στην ε, ίδια τη χώρα. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματική δέσμευση από πλευρά όλων. Ειλικρινής δέσμευση για να οδεύσουμε προ την ειρήνη και να αποδεχτούν ότι μόνο η πολιτική επίλυση θα μας οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ε, νομίζω ότι Ακόμη σήμερα κάποιοι από τους εταίρους μας στο επίπεδο της διεθνής κοινότητας δεν έχουν πιστεί για την πορεία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ευχαριστήσω το σύνολο των ε, προστεκλημένων μας, το σύνολο των ε, παρεμβενόντων, οι οποίοι ήρθαν ως εδώ και μας παρουσίασαν την ε, τόσο εντυπωσιακή εργασία που πραγματοποιείται καθημερινά και όλοι μπορέσαμε να έχουμε μια απτή εικόνα του πώς έχει η κατάσταση σήμερα, πόσο ε, ε, είναι δραματική και πόσο 6 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια και από την ε, συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλους και να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Προβέρα, για να ολοκληρωθεί η κοινή συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και μας βοήθησε να σκεφτούμε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα εκεί. Και πάλι ευχαριστώ.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

ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα, εφόσον δεν σας ενδιαφέρει το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε και το οποίο έχει να κάνει με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. No interview, no, no, no, no. Can you do that outside, please?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 Φτάνουμε στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ προβλέπεται ανταλλαγή απόψε σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προφορικής ερώτησης με τελικό ψήφισμα. 45 λεπτά παρακαλώ. συζητάμε με το ελεγκτικό συνέδριο για την ειδική έκθεση Σεπτεμβρίου, πράγμα το οποίο θα δώσει τροφή στη σκέψη μας για να καταλήξουμε σε τελικό ψήφισμα. Είναι η τιμή που έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Βέσπερκ, που είναι μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, που έχει εκπονήσει και την ειδική αυτή έκθεση για την διακυβέρνηση στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουν μείνει πολύ τέλος πάντων. Το λεκτικό συνέδριο με την έκθεσή του δεν φαίνεται πολύ ευχαριστημένο όσον αφορά την διαχείριση της αρρωγής μας στη μεγάλη αυτή χώρα η οποία είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους αλλά πολύ φτωχή όσον αφορά το καθάριστο εθνικό προϊόν. Έχετε πει ότι η στρατιωτική κατάσταση και η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια επί τόπου, ιδίως ανατολικά και στα δύο κύβου, έχει οδηγηθεί σε αλλαγές με την νίκη των στρατικών δυνάμων και της Μινόσκου επί της M3. Παραμένουν βέβαια μεγάλες αβεβαιότητες. Η προτεραιότητα είναι η ειρήνευση, η εξουδέρωση των άλλων ένοπλων δυνάμεων που για καιρό κυριαρχούν στην περιοχή. Υπάρχουν μέσα για να βελτιωθεί λοιπόν η διακυβέρνηση στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό με χρηματική βοήθεια αλλά και με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών. Ο ειδικό μας απεσταλμένος επίσης στη περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ο κύριος Φερβάκε μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν κάποια μικρή ακτίδα αισιοδοξία για την χώρα αυτή αλλά επειδή τα ιστορικά δεδομένα είναι αυτά που ξέρουμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για κάθε πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τη βοήθειά μας σε αυτή τη χώρα. Συνεπώς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσουμε την ειδική έκθεση που έχετε να μας παρουσιάσετε κύριε Βέσπερκ. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα το να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση σε σχέση με, ε, τον λογιστικό έλεγχο της ε, βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταρρυθμίσεις και τη δημοκρατικοποίηση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Γιατί κάναμε μια τέτοια μελέτη για, την, για το εύθραυστο ενός κράτους. Η καλή διακυβέρνηση είναι βασικός γνώμονας της επιτυχίας μιας ε, αναπτυξιακής βοήθειας και βοήθειας για τη δημοκρατικοποίηση. Αυτή τη στιγμή όμως περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άτομα ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και σε κράτη που έχουν αστοχήσει. Παρά τις ε, σημαντικές προσπάθειες και τις ε, δεσμεύσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη βοήθεια που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένη η αξία αυτής της βοήθειας σε σχέση με το κόστος τους. Οι χώρες αυτές απέχουν ακόμα περισσότερο από τις άλλες σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Το συμπέρασμά μας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε έναν των κρατών που βρίσκονται σε κατάρρευση των κρατών που έχουν αστοχήσει πρέπει να μεταρρυθμιστεί η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους της και κατά πόσο είναι αποτελεσματική. Η έρευνά μας κάλυψε 16 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κύριους τομείς διακυβέρνησης, τη διαδικασία εκλογών, ε, ο τομέας ασφάλειας, αποκέντρωση και άλλα θέματα στο χρονικό διάστημα 2003-2011. Ο το συνολικό κόστος αυτών των προγραμμάτων έφτανε στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι εμείς ελέγξαμε ένα μείγμα παλαιότερων και νεωτέρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πόσο ήταν η απόδοση αυτών των προγραμμάτων μέσα στον χρόνο. Επελέγει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ως αντιπροσωπευτικό δείγμα γιατί θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο εύθραυστα κράτη στον κόσμο και λόγω του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος, ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς εταίρους της με χρηματοδότηση 1,9 δισεκατομμυρίων στο χρονικό διάστημα 2003-2011. Ενώ η Κομισιόν και η Υπηρεσία εξωτερική δράση είχαν θεσπίσει πλήρη, μια πλήρη στρατηγική δράση που καλύπτανε και τον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα και τον τομέα ασφάλειας για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις σε επίπεδο μεμονωμένων προγραμμάτων. Λιγότερο από μισά από τα προγράμματα έδωσαν καρπούς ή είναι πιθανότητα ε, <clears throat> πιθανότητα δώσουν καρπούς σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Η πρόοδος στο διάστημα που καλύπτει η ερευνά μας ήταν περιορισμένη και γενικά χωρίς να επιτύχει τους περισσότερους στόχους της η βιωσιμότητα των προγραμμάτων αυτών δεν φαίνεται να είναι ρεαλιστικός στόχος. Λόγω του έφθος του πλαισίου μπορούν να κατανοηθούν πολλά από αυτά τα γεγονότα, αλλά η έρευνά μας είδε και περιπτώσεις όπου η ίδια η σχεδίαση των προγραμμάτων και οι ασαφείς στόχοι καθώς και η ανεπαρκής διαχείριση του κινδύνου έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποτυχία των προγραμμάτων αυτών. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν έχει χρησιμοποιήσει επαρκώς την ερεσιμότητα ε, για να προωθήσει ορισμένα προγράμματα προτού ξεκινήσουν ή προτού συνεχίσει η χρηματοδότησή τους. Είναι σύστασή μας ότι ακολουθώντας το θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας προς κράτη που έχουν αστοχήσει, η Κομισιόν να εξετάσει τα εξή μέτρα για να βελτιωθεί η σωστή, η σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, η Κομισιόν και η Υπηρεσία εξωτερική δράση θα πρέπει να επαναξετάσει τη γεωγραφική κατανομή της βοήθειας στις επαρχίες του Κονγκό και να δώσει περισσότερη έμφαση στο να υπάρξει καλύτερη λογοδοσία σε σχέση με τη διακυβέρνηση στο Κονγκό. Δεύτερον, όταν αναλαμβάνει τον κίνδυνο της παρουσίας της η Κομισιόν θα πρέπει να έχει πιο οξυμένη αξιολόγηση κινδύνου για να μπορέσει να υπάρχει καλύτερη στοχοθεσία εν ώψη της περιορισμένης δυνατότητας εφαρμογής και απορρόφησης των κονδυλίων. <clears throat> Λαμβάνοντα υπόψη δηλαδή την διαφθορά, την αδυναμία της ε, τοπικής διοίκησης, την έλλειψη δυνατοτήτων παρακολούθησης κτλ. Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο η Κομισιόν θα πρέπει να βρει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των στόχων της και του εφικτού ρεαλιστικά. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει και μια εσωτερική εθνική δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους κύριους εταίρους του Κονγκό. Πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης και των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί σε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κονγκό. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να ελεγχθεί η συμμόρφωση με αυτούς τους στόχους, όπου υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων και δράσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει εγκαίρως και αναλογικά όταν αυτό απαιτείται. Τέλος, ο πολιτικός διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κονγκό θα πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να είναι πιο απαιτητικό, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανόηση να γίνεται έγκαιρα και να γίνεται με τους κατάλληλους τρόπους. Εάν ακολουθηθεί λοιπόν αυτή η σειρά κριτηρίων, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματική η βοήθειά μας και να οδηγήσει ταχύτερα σε μια συμφωνία σε σχέση με τις προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τους στόχους και τους κινδύνους του προγράμματος. Κάτι το οποίο θεμελιώθηκε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποδίδει καρπούς με τη μορφή μεταρρυθμίσεων. Για να κλείσω. Η έκθεση αυτή έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή γιατί η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι έτοιμη να οριστικοποιήσει το πλαίσιο σχέσεων με το Κονγκό για το, τη χρηματοδότηση το χρονικό διάστημα 2014-2020. Αυτές λοιπόν οι συστάσεις έρχονται στην κατάλληλη στιγμή να βοηθήσουν την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βάισπέργια. Θα έπρεπε να, να δώσουμε το λόγο στον Μπάς ο οποίος είναι ο εισηγητής για αυτή την έκθεση. Κυρία Σαρζεντίνη, μπορείτε να παίξετε το ρόλο του Μπάς Όχι. Μπορείτε να τον αντικαταστήσετε. Ούτε. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Βέισπεργκερ. πόσο σας ικανοποίησε όσα ακούστηκαν, πόσο σας όσα ακούστηκαν στον τύπο από, μετά την ε, δημοσίευση της εκθεσής σας. Τα σχόλια στον τύπο ήταν τόσο σκληρά που μετά οι ενημερώσεις μας ήρθαν ε, και η αποδελτίωση ε, ανέφερε 9 δις που διασπαθίστηκαν στη Δημοκρατία του Κονγκό. Εσείς τώρα δηλώνετε κάτι ακόμη πιο ε, εντυπωσιακό, επίκαιρο αυτό που λέτε για την ανάγκη προσαρμογών και βελτιώσεων της χρηματοδότησης και για λογοδοσία της χρηματοδότησης στην Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες χώρες. Αυτή είναι μια συζήτηση που θέλετε να ξεκινήσει εδώ, αλλά εσείς πόσο χαρήκατε με τα δημοσιεύματα στον τύπο και τα αποτελέσματα που ανέφεραν. Πρόεδρε, μου ζητάτε ουσιαστικά να κάνω έλεγχο στον ελεύθερο τύπο. Στην τυπία δεν είναι αυτό όμω αρμοδιότητα του ελεγκτικού συνεδρίου να επισημάνω ότι ο τύπος είναι τύπος. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που είναι. Κάποιες φορές έχουν ε, την τάση να ε, βάλουν κατά των πλέον ενδιαφερόντων και κυρίως με πρωτοσέλιδα. Δεν αναγνώριζα αυτά που διάβαζα στα πρωτοσέλιδα σε σχέση με το περιεχόμενο τη εκθεσή μου και δεν θα κάνω εγώ έλεγχο στον ελεύθερο τύπο. Πρόεδρο. Νομίζετε όμω ότι τα δημοσιεύματα στον τύπο και ο τόνο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτά και οι διατυπώσεις εκάλυπταν επαρκώ και ικανοποιητικό στο περιεχόμενο τη έκθεση. Ναι. Εγώ όχι. Οπότε προφανώς διαφωνούμε. Είμαι πρώην δημοσιογράφος και είμαι και πολιτικός ε, άνδρας. Μέχρι πριν λίγους μήνες ήμουν. Να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την ε, σημασία του τύπου, αλλά και το κατά πόσο είναι ακριβά, ακριβή τα δημοσιεύματα στον τύπο. Ο λόγος τώρα στον κύριο Κάρπεντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, οι παρατηρήσεις μου θα συμπληρωθούν από τον κύριο Χάμερτατ από την Επιτροπή, αλλά μερικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και εμείς διαβάσαμε τα δημοσιεύματα στον τύπο για την έκθεση, έχουμε τις δικές μας απόψεις, όμως πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δικό μας το ρόλο στη διαδικασία προγραμματισμού. Κυρίως το τι θα γίνει στο μέλλον και πώς θα ε, ε, υλοποιήσουμε τις αρχές που προκύπτουν από την έκθεση. Το πρώτο είναι η πολλαπλή διαχείριση του κινδύνου. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στην Κινσάσα σε μια κοινή αποστολή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος πλαίσιο για την δημοκρατία του Κονγκό. Είδαμε τι πολιτικές απειλές υπάρχουν στη χώρα λόγω του έθραυστου περιβάλλοντος. Είδαμε τα επιχειρησιακά προβλήματα και το θέμα του δικαστικού τομέα αυτό νομίζω καλώς έχει υπογραμμιστεί σε πολλές σχετικές μελέτες για το εύθραυστο περιβάλλον. Το ευάλωτο αυτό περιβάλλον, το επισφαλές περιβάλλον που δημιουργείται και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια και προβλεψιμότητα στη χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Η προστασία των φορέων, η τήρηση των κυβερνητικών ε, δεσμεύσεων στα πλαίσια της λογοδοσίας επίσης και αυτό είναι μια από τις ε, πηγές του αποτελεσματικού κυβερνητικού διαλόγου, κάτι που τόνισε ο κ. Βάισπερκερ. Και επίσης ο σωστός σχεδιασμός των προγραμμάτων και των project είναι, πρέπει να είναι ρεαλιστική η στόχη αλλά και φιλόδοξη κάποιες φορές. Να πω δύο λόγια και για το πολιτικό τοπίο, διότι τέθηκε το θέμα της γεωγραφικής κατανομής της χρηματοδότησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει δίκαιη γεωγραφική κατανομή σε τομεί όπω η υγεία και η περίθαλψη. Το συζητήσαμε και με άλλου αναπτυξιακού μεσαιτέρου στην Κινσάσα για το πού θα δραστηριοποιηθούν εκείνοι και πού εμεί, λαμβάνοντα υπόψη το ιστορικό που έχουμε σε αυτή την τόσο εκτεταμένη χώρα. Επίση, οι πολιτικέ συνέπειε είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τη Καμπάλα, όπου αναφερθήκατε κι εσεί ο ίδιο. Εδώ Μιλάμε για μια πολύ σημαντική σειρά από ευκαιρίες, όχι μόνο για την βόρειο-ανατολική δημοκρατία του Κονγκό, εκεί υπάρχει διεθνής ρόλος που πρέπει να αναλυφθεί ούτως ή άλλως, αλλά μπορεί να είναι και αποτελεσματική η παρέμβαση. Επίσης, δύο ακόμη σχόλια. Πρώτον, εργαζόμαστε μετά την πρόσφατη επίσκεψή μα για να υπάρχουν συγκεκριμένε κυβερνητικέ δεσμεύσει ε, σε όλου του τομείς που μα ενδιαφέρουν. Μιλήσαμε στα υπεύθυνα υπουργεία, του υπουργού και του ανώτατου αξιωματούχου. Αυτό είναι το σωστό σημείο αφετηρία για να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση στη χώρα. Και έπειτα πιστεύουμε Είμαστε πεπισμένοι ότι οι παρεμβάσει στου ε, τομεί προτεραιότητα θα πρέπει να συνοδεύονται από, τα εύστοχα, από εύστοχα μέτρα στον τομέα τη σωστή διαχείριση με σωστή αλληλουχία, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, η αιρεσιμότητα, κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένω, είναι σημαντικό να τονίζουμε διαρκώς ότι εδώ λειτουργούμε στο πλαίσιο των συμφωνιών του Ιθικοτονού. Δηλαδή, μια προσέγγιση που βασίζεται στον πολιτικό διάλογο και την εταιρική σχέση και συνεργασία. Οι σχέσεις μας με τη δημοκρατία του Κονγκό θεμελιώνονται σε μια σειρά από διεθνείς αρχές που έχουν να κάνουν με την αμοιβαία λογοδοσία, τη νέα συμφωνία και το καθεξής. Νομίζω πάντως ότι το πολιτικό σκηνικό που ισχύει, το πολιτικό περιεχόμενο που ισχύει για τις χώρες ΑΚΕ ισχύει και εδώ. Κύριε Κάρπεντερ, η έκθεση κάνει λόγο και για τους χιλιάδες αστυνομικούς που εκπαιδεύτηκαν. Και προφανώς κανείς δεν λογοδότησε για αυτούς. Δεν έχει εξελιχθεί το πρόβλημα. Αλλά πού πήγαν, τι απέγιναν. Έχετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε ότι ήταν κάπως παράξενο αυτό το στοιχείο. Δεν θέλω να υπεκφύγω, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την εκτέλεση του προγράμματος. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, συμμετείχαμε σε μια σειρά από δράσεις για να στηρίξουμε τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας στο αστυνομικό κλάδο. ιδίω μετά από την ε, αποστολή της EUPOL στη δημοκρατία του Κόγκο. Είδαμε μετά την επίσκεψη αυτή ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ακριβώς αυτή η μεταρρύθμιση. Θα χρειαστεί να υπάρξει μεταρρύθμιση ολόκληρου του τομέα ασφαλείας με ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση και όχι έξωθεν προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα και διαρκή αποτελέσματα. θα πρέπει η κατάρτιση των αστυνομικών να συνεχιστεί σε προσωπικό επίπεδο. Ξέρουμε λοιπόν που βρίσκονται στη χώρα, ξέρουμε τι κάνουν και ξέρουμε τι έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν. Δεν μπορεί κανείς να επινοήσει εκ νέου την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την αποτελεσματική πολιτική κατάρτιση και την αποτελεσματική κατανομή πόρων. Δεν μπορεί κανεί να τα ε, επινοήσει εκ νέου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικέ οι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώ σε αυτέ. Ερχόμαστε τώρα στον Κιάρα Μιλάν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέτω λόγο. Σας ευχαριστώ. Πιέρα Μιάντ, είμαι διευθυντής της ΕΦΚΟ για την ε, Δυτική Αφρική και την Κεντρική Αφρική. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία, διότι εμείς είμαστε, όπως είπε ο συναδελφός μου, ε, υπεύθυνοι για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, για να πούμε ότι παντού υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ε, κατάρτισης οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια εκπαίδευση με κατάρτιση φεύγουν από τη διοίκηση, πηγαίνουν σε άλλες δουλειές. Κάτι το πολύ φυσιολογικό. Αυτό το οποίο έγινε στην πραγματικότητα ήταν ότι υπήρξε μια μονάδα ειδική αστυνομία η οποία καταρτίστηκε για να προστατεύσει τις εκλογές και μετά από τις εκλογές διαλύθηκε αυτό το, αυτή η μονάδα αλλά αυτοί οι αστυνομικοί βρίσκονται σε άλλες μονάδες αν το δούμε απλώς σαν ένα θέμα κατάρτισης, η κατάρτιση αυτή δεν πήγε στράφη, απλώς τα άτομα αυτά τα οποία έλαβαν αυτή την κατάρτιση δεν βρίσκονται πια μαζί σε μια ειδική μονάδα η οποία δημιουργήθηκε με την ευκαιρία των εκλογών και έχουν περάσει σε άλλες μονάδες, δεν έχουν εξαφανιστεί στο δάσος λοιπόν. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε και να εκπαιδεύουμε την αστυνομία στο Κονγκό ιδίως σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αστυνομικών αρχών, ώστε αυτή η υπηρεσία να γίνει πιο επαγγελματική και να ξέρουμε πράγματι ποιος είναι αστυνομικός και ποιος θα πρέπει επομένως να αμείβεται. Να κάνω και κάποια σχόλια τώρα σε σχέση με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, αν μου επιτρέπετε, και θα ήθελα να πω όπως είπε η κυρία Άστον και ο κύριος Φίμπαξ στο παρελθόν ενώπιον του ε, Ελεκτικού συνεδρίου. Λαμβάνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τις ε, συστάσεις του Ελεκτικού συνεδρίου κάθε φορά που αυτό μας οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής ανάπτυξης ιδιαίτερος. Χαίρομαστε πάρα πολύ που μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιες συστάσεις. Του του λεχθέντος όμως θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που αναφέρθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο. Ελέγχθη ότι <clears throat> είναι ένα υπόδειγμα κατά κάποιο τρόπο ευάλωτου κράτους η δημοκρατία του Κονγκό. Ένα παράδειγμα που μας επιτρέπει να αντλήσουμε γενικά συμπεράσματα για το σύνολο των κρατών που βρισκόνται σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Στην περιοχή που με ενδιαφέρει εμένα, που είμαι αρμόδιος, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κρατών σε κατάσταση τρωτή και πρέπει να σας πω είναι πολύ δύσκολο να γενικεύσει κανείς την κατάσταση αυτών των κρατών. Υπάρχουν ορισμένε αρχές ε, ε, για τα κράτη αυτά και αυτό κάναμε στην Μπουζάν όταν έγινε το λεγόμενο New Deal αλλά δεν μπορεί να μεταφέρει κανείς μηχανιστικά συμπεράσματα που αφορούν μια χώρα σε άλλες χώρες, παραγωγός χάρη από το Κονγκό στο Μαλί και αντιμετωπίζοντας άλλες χώρες όπως είναι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο εύθραυστες αλλά δεν έχουν εμφανιστεί τόσο πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί <clears throat> όταν θέλουμε να καταλήξουμε με ένα περιορισμένο ε, δείγμα σχέδιων, ορισμένα από τα οποία ήταν ακριβώς στο στάδιο κίνησης όπως ελέγχθη πολύ σωστά. Δεν μπορούμε από όλα αυτά να αντλήσουμε γενικότερα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις για τα στα κράτη. Μία από τις ε, μομφές που μας ε, απευθύνει το Ελεκτικό συνέδριο είναι η υπερβολική φιλοδοξία στα προγραμματά μας και η έλλειψη ρεαλισμού που είναι η άλλη όψη του νομίσματος της φιλοδοξίας. Μιλάμε εμείς για τα θέματα της ε, ευκυβερνησίας, υποστήριξη στη δικαιοσύνη, στην εκλογική διαδικασία, αυτά και τα θέματα που κοίταξε το ελεκτικό συνέδριο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σχέδια που αντανακλούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε αξίε προσαρμοσμένε μέσα εισαγωγικά σε κάθε χώρα. Για τι εκλογέ, παραδείγματο χάρη, όταν εμεί ξεκινάμε ένα σχέδιο, δεν θα αρχίσουμε να λέμε, να σκεφτόμαστε ότι οι εκλογέ οι οποίε θα προκύψουν θα είναι κατά το ίμιση μονάχα ή κατά 25% μονάχα δίκαιε και αμερόληπτε. Όχι, ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να είναι απόλυτα αμερόληπτε και δίκαιε αυτέ οι εκλογέ και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Το να μας ψέξει κανείς στη συνέχεια ότι είχαμε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους, εντάξει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να επανέλθω, η γεωγραφική κατανομή των σχεδίων, πολύ σωστά απήντησε ο συνάδελφό μου από τη διπλωματική υπηρεσία. Φυσικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το έδαφο μια χώρα. Αλλά είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη δεν μπορεί να τον πράξει αυτό. Και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να μπορέσουμε να κατακαιρματίσουμε τόσο πολύ τις ενεργειές μας αν θέλουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ένα θέμα αποτελεσματικότητος, συνεργασίας <clears throat> με τους άλλους εταίρους που δρούν στη δημοκρατία του Κονγκό για να μπορέσουμε να έχουμε κατανομή αρμοδιοτήτων και γεωγραφική κατανομή. Αυτό είναι θέμα διακυβερνητικών συμφωνιών για το πώς θα λειτουργήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο και τέλος θέλω να πω ότι στο ένατο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης θα υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των προσπαθειών μας στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό. Εκεί υπάρχει μια γενικότερη συνένεση. Υπάρχει η προσπάθεια των ΗΠΑ και της Μέρι Ρόμπινσον συγκεκριμένα που πρέπει να υποστηριχθεί για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρεται σε έλλειψη συμμετοχής και πρωτοβουλίας από την πλευρά του, της κυβέρνησης του Κονγκό. Οι συναδελφοί μου που επανέρχονται από την, από και ήταν προηγουμένως στο Κονγκό, είπαν ότι το, πρώτο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν αφού επισκέπτηκαν μαζί με τους συναδέλφους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ορισμένα Υπουργεία, υπάρχει έλλειψη συνομιλητών, έλλειψη θέλησης, ανάληψης τις ευθύνης για αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και αυτό είναι δυσμενές γιατί εκεί βρίσκεται η εστίαση της προσπάθειάς μας να υπάρξει τοπική ανάληψη ευθύνης για όλα αυτά τα προγράμματα. Κλείνω τώρα με κάτι άλλο το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό από μεθοδολογική άποψη θέμα και πρόκειται για την χρήση της αιρεσιμότητας <clears throat> και ακόμα και της προαιρεσιμότητας για τη βοηθεία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί αυτό είναι μια μορφή προσέγγισης της βοήθειας αναπτυξιακού χαρακτήρα και για μας, όπως ελέγχθη από τον συνάδελφό μας προηγουμένως, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία με μια κυβέρνηση επί τη βάση διαλόγου για κοινού στόχους και δεν πρόκειται καθόλου για μονομερή επιβολή συνθήκων και ερεσιμότητας και προερεσιμότητας για τον τρόπο εργασίας. Σε επίπεδο εφαρμογής των σχεδίων εμείς το έχουμε κάνει αυτό επί τη βάση της εταιρικής σχέσης της Κοτονού. Δεν μπορεί να υπάρξει μηχανισμός ο οποίος να ενσωματώνεται σε κάθε σχέδιο που να καταλήγει σε μία μόνιμη εκκίνηση και μετά ε, ανάσχεση. Δεν μπορούμε να έχουμε γραφειοκρατική λειτουργία που να οδηγεί σε αυτόματη ανάσχεση των προγραμμάτων επειδή δεν τηρήθηκε κάποιος όρος. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να έχουν μια τέτοια απόλυτη αιρεσιμότητα αλλά θα πρέπει να σας πω ότι η δική μας εμπειρία <clears throat> σε πάρα πολλά σχέδια έδειξε ότι μια τέτοια δράση είναι καταστροφικού χαρακτήρα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα, αλλά η αιρεσιμότητα πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα και η κρίση η οποία γίνεται από τους εταίρους της Δημοκρατίας του Κονγκό να είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Για παράδειγμα, εμείς υποστηρίζουμε τη διενέργεια των εκλογών. Είναι ένα πραγματικό λοιπόν παράδειγμα η κυβέρνηση του Κονγκό αποφασίζει να αλλάξει το Σύνταγμα μέσα στην εκλογική διαδικασία. Κάτι πολύ κακό. Τι σημαίνει αυτό. Σταματάμε τη βοήθεια για τι εκλογέ με κίνδυνο να μην γίνουν καθόλου εκλογέ ή συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε. Όταν λέω ότι αντιμετωπίσαμε εμεί, είναι όλο ο κόσμο τελικά. Όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και να το δίλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και κλείνω εδώ. Πρέπει να πω ότι είναι κρίμα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί από τη μια πιστεύω ότι το λεκτικό συνέδριο εξέδωσε μια πολύ ισχυρή και σε βάθος έκθεση, από την άλλη, πολύ σωστά λέτε ότι η αιρεσιμότητα υπό τη στενή έννοια του όρου οδηγεί σε καταστροφή των αναπτυξιακών σχέσεων. Αν ε, ερμηνεύω σωστά ερμηνεύοντας ελεύθερα κάπως αυτά που είπατε. Πάντως τελικά είναι ο φορολογούμενος, ο οποίος απαιτεί να δει που πάνε τα χρήματά του και ότι πιάνουν τόπο. Συνεπώς το ελεκτικό συνέδριο δεν πρέπει να κοιτάξει μόνο την δημοσιονομική πτυχή, αλλά να δει και την απόδοση των πολιτικών μας. Συνεπώς, κατά την άποψή σας, εδώ η έκθεσή σας σπρώχνει προς μια πιο αυστηρή ρεσιμότητα από αυτήν που εσείς θεωρείτε επιθυμητή από πλευράς αναπτυξιακών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της, σωστά. Ναι. Είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση. Γιατί ακούγεται σαν είμαστε κατά, αλλά δεν είμαστε κατά είμαστε κατά μιας μηχανικής προσέγγισης που απαιτεί αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να είναι μονομερές αυτό, πρέπει να είναι κάτι που θα έχει συμφωνηθεί. Είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Τότε μόνο υπάρχει η νομιμότητα. Αυτή είναι η νέα ιδέα. Πρέπει δηλαδή τους στόχους να τους ενστερνίζεται η κυβέρνηση που έχουμε απέναντί μας. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να λειτουργούμε μόνο μηχανιστικά, βάσει ενός εγγράφου δηλαδή δεσμευτικού, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας και ότι το αποτέλεσμα των κυρώσεων σε εισαγωγικά ή τέλο πάντων της διακοπής, της αρρωγής μας, ε, συγχρόνως πρέπει να συνοδεύεται από την πολιτική οπτική γωνία για να δούμε δηλαδή τι συνέπειες θα έχουν αυτές οι εντό εισαγωγικών ε, κυρώσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο βέβαια λειτουργεί μέσα σε κάποια περιθώρια βεβαιότητας. Παρακαλώ κύριε Βεσμπερκ, τελευταίος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ ότι είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι μια από τις πιο σημαντικές συζητήσεις που έχουμε τελευταία. Η αιρεσιμότητα πιστεύω εγώ ότι πρέπει να συζητηθεί παρατέρω και ο ε, από την Κομισιόν και εγώ συμφωνούμε ότι είναι σημαντική αιρεσιμότητα. Από την άλλη μεριά όμω δεν καταφέρουμε να δούμε την αιρεσιμότητα και στα πλαίσια της απόδοσης. Δεν θέλω να μπω περισσότερες λεπτομέρειες τώρα, αλλά πάντως θέλω να υπογραμμίσω ότι η ίδια η Κομισιόν δεν έκανε μια από τις τελευταίες πληρωμές σε σχέση με τις εκλογές. Να, κάποιο είδου αιρεσιμότητα. Κατά πόσο τώρα είναι πολιτικού χαρακτήρα ή έχει να κάνει με τις επιδόσεις δεν ξέρω. Πρόεδρος, πραγματικά θα ήθελα κύριε Βέσμπερ, εσείς και ο κύριος Σπίγκστον που έκανε την έκθεση για την Αίγυπτο και εσείς για την Παλαιστίνη, όλοι μαζί... Α, εσείς, ωραία να βρεθούμε μαζί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να λύσουμε τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Εσείς έχετε αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντα αυτά του ελέγχου της απόδοσης. Εδώ τίθενται πολλά πολιτικά ζητήματα, όπως βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι αναπόφευκτα. Πολύ θα θέλαμε λοιπόν να μπούμε περισσότερο σε βάθος από ό,τι σήμερα. Πάντως η Αναπτυξιακή Επιτροπή να ξέρετε ότι θα τα παρακολουθεί όλα αυτά στενά. Η Εύα Ζολή τώρα. Μέχρι τώρα την αντικαθιστούσα εγώ απλώς. Παρακαλώ. nous avons une transition toute... Ωραία. Μετά τον έλεγχο του λεκτικού συνεδρίου της βοηθειάς μας προς το Κονγκό και το σημείο 19, η αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ασταθή κράτη, μας επαναφέρει στη σειρά των εργασιών μας. Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι εδώ εκ μέρους της Επιτροπής μας τους δύο συντάκτες της μελέτης που εξετάζουμε σήμερα για τα θέματα τα οποία διακυδεύονται όσον αφορά τις πιο ευάλωτες χώρες. Είναι η κυρία Μικάελα Κάβας και ο κύριος ε, Edward από την Overseas Development Institute του Λονδίνου. Κυρίες και κύριοι, Έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τα κύρια σημεία της μελέτης σας, παρακαλώ. Οι ευρωβουλευτές μετά μπορούν να πάρουν το λόγο. Και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσετε, να αντιδράσετε. Η κυρία Μικαέλα Γαβάς πρώτα. Και μετά ο κύριος Έντουαρτ. Με τη σειρά που θέλετε βέβαια. Καλησπέρα σας. Είμαι από το υπερπόντιο ίδρυμα για την ανάπτυξη, το ODI, στο Λονδίνο, και να πω ότι η έκθεση που ετοιμάσαμε μιλά για την, για την κατάσταση της αναπτυξιακής βοήθειας και τις σχετικές προκλήσεις. Παραγγέλθηκε τον Απρίλιο του 2013 περίπου. Ξέρουμε ότι από τότε έχουν προκύψει εξελίξεις και η παρουσίαση μας σκοπό έχει να καλύψει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις ενώ βλέπετε την παρουσία στην οθόνη σας, θα ήθελα να θυμάστε ότι είναι τέσσερα τα βασικά μηνύματα που προσπαθώ να μεταδώσω. Πρώτα απ' όλα την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ευάλωτα κράτη. Έπειτα η συνοχή στη δράση των διαφορών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και το κατά πόσον καταφέρνουν να λάβουν υπόψη σωστά τις προκλήσεις των βάλωτων ε, κρατών. Εδώ είχαμε αρκετά επικριτικά σχόλια. Έπειτα το είδος των ε, μέσων ή τέλος πάντων των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται και εδώ πραγματικά μας εξέπληξε η τελο παντων των διαδικασιων που χρησιμοποιουνται και εδω πραγματικα μας εξεπληξε η προκληση του πώς να περάσουμε από την ανθρωπιστική σκοπιά στην αναπτυξιακή δηλαδή από την κάλυψη των κατεπηγουσών αναγκών, στο πώς θα αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμες και θεσμικές ανάγκες. Πρώτον, λοιπόν, δυνατότητες. Υπήρχε μια σειρά από προκλήσεις, μια σειρά από απαιτήσει εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό το πλαίσιο και μας απασχόλησε κατά πόσον υπήρχαν σωστές δεξιοτεχνίες συνδυασμένες με τις, απαραίτητε, με τις ε, επιδιωκόμενες ανάγκες προσκάλυψη και στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Επικεντρωθήκαμε στην πρόληψη, τέλος πάντων την ε, προηγούμενη φάση από την παρέμβαση. Περνάω τώρα στην ίδια μου την παρουσίαση, θα την ε, σχολιάσω πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο της, των ευάλωτων κρατών. Μετά ο συνάδελφος θα σχολιάσει τα συγκεκριμένα πορίσματα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το τοπίο της ένδυας μεταβάλλεται και συνεχίζει να μεταβάλλεται. Τα δεδομένα αυτά είναι κοινότοπα πλέον. Αλλά είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος των φτωχών ζουν πλέον σε κράτη ευάλωτα. Μια από τις μεγαλύτερες λοιπόν προκλήσεις είναι να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτήν την ευάλωτη φύση των κρατών μαζί με τη φτώχεια που δεν είναι θέματα διακριτά. Να θυμηθούμε ότι ευάλωτα κράτη δεν μπορούν να πετύχουν συνήθως τους στόχους της χιλιετίας και έτσι χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα. Και κάποιες χώρες αυτές της πρώτης ομάδας δεν έχουν καταφέρει κανένα από τους στόχους της χιλιετίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί για τα ευάλωτα κράτη, ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν, τα φαινόμενα βίας, το ξέσπασμα βίας και το πώς επιδεινώνει τη λειτουργία των θεσμών είναι κάτι το εντυπωσιακό που πρέπει, και πρέπει να μελετηθεί κανείς, να μελετηθεί γενικώ. Ε, τι γίνεται τώρα με τον κατάλογο των ευαλωτών κρατών. Διαρκώς εξελίσσεται ο κατάλογος αυτός αλλά βλέπετε ότι είναι ανάμεκτη η ομάδα αυτή των χωρών. Είναι αρκετά πολύ πίκυλη. Από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από αρκετές χώρες βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να αλλάξουν κατηγορία. Τώρα, η φύση της χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποιες βασικές συνιστώσεις που επαναλαμβάνονται στη χρηματοδότηση. Στοιχεία του 2010 από τον ΩΣΑ σε αμερικανικές από την αμερικανική πλευρά βλέπουμε το μεγαλύτερο δωρητή προς τα ευάλωτα κράτη, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν επίσης σημαντικό ρόλο για την αναπτυξιακή βοήθεια 50 δις ε, συνολικά, 50 δις δολάρια και ένα μέρος από αυτήν είναι βασισμένο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Το μεγαλύτερο μέρος μάλιστα των ποσών αυτών απευθύνονται σε 7 χώρες, πέραν όλων των υπολείπων που είδατε στον κατάλογο. Κονγκό. Είναι είδος χώρα στο Κονγκό, τυπολογία χώρας, ε, χώρες που συνήθως εξαρτώνται από έναν και μόνο δωρητή. Το αντίστροφο Αντίστοιχη κατάσταση όμως είναι η πραγματική πρόκληση. Κάποιες από τις αρχές τώρα, από τις αρχές που όλοι έχουμε αποδεχτεί, βάσει των καλών πρακτικών σε αυτό το πλαίσιο. Ένας βασικός στόχος είναι η οικοδόμηση του κράτους. Το κατά πόσον δίδεται έμφαση στα μέτρα πρόληψης το κατά πόσον αναγνωρίζονται οι συσχετισμοί μεταξύ των πολιτικών στόχων και των κοινωνικών. Θα πρέπει στα ευάλωτα κράτη να γίνεται αξιολόγηση όλων των στόχων και όλων των διαδικασιών. Η μη διακριτική μεταχείριση, η συμμετοχή στην κοινωνία προκειμένου να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση προς την σύγκρουση. Οι μηχανισμοί συντονισμού, οι τοπικές προτεραιότητες, οι ταχύτητα αλλά και η επιμονή. Δεν μπορεί κανείς να κάνει συνεχώς έναν αγώνα δρόμου ή μαραθώνιο. Πολλές φορές χρειάζεται εναλλαγή όμως ή ταυτόχρονη πορεία και των δύο δρομέων για την οικοδόμηση των θεσμών. Επίσης η αποφυγή του αποκλεισμού, των θυλάκων αποκλεισμού είναι και αυτό σημαντικό. Η μελέτη εξήβρε ότι σταδιακά οι περισσότεροι φορείς βοήθειας δεν έχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ιδιαίτερες προκλήσεις των ευαρατών καταστάσεων, ακόμη παρά τις ε, εντυπωσιακές τους δεσμεύσεις πολλές φορές. Περνάμε τώρα στα πορίσματα των επιδόσεων σε σχέση με όλα αυτά. Ένας κατάλογος δείχνει τις βασικές τις προκλήσεις Κάτι που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το εθνικό ε, τοπίο. Και το, επίσης το πόσο καλά συντονισμένες είναι οι διεθνείς προσπάθειες. Κάποιες φορές υπάρχουν βλαβερές συνέπειες, αφαρά τόσο περίπλοκα και βάλα τα περιβάλλοντα. Ο κατάλογος είναι πολλές φορές μια καλή εικόνα των αρνητικών επιπτώσεων. Ένα άλλο ζήτημα το βλέπετε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Η νέα συμφωνία για δέσμευση υπέρ των ευάλωτων κρατών. G7 G7-SIN. 18 ευάλωτα κράτη είχαν οριστεί το 2011 στο Αμπισάν και δεν μας απασχολεί μόνο η πλευρά της παροχής βοήθειας, αλλά και της προσφοράς, της ζήτησης μάλλον. Πάντως, υπάρχουν κάποιες χώρες που διαρκώς επανέρχονται στον κατάρτιση προτεραιοτήτων τους για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Εδώ πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες του ευάλωτου χαρακτήρα, κάτι που καταλήγει σε πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των κρατών αυτών. Επίσης, οι εθνικοί φορείς, κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών, ε, πολίτες είναι οι πλέον αρμόδιοι για να ε, δώσουν εξηγήσει για τον ευάλωτο χαρακτήρα του κράτους τους και το για το τι ανάγκες που να καλύπτουν τα προγράμματα. Τρίτον, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνήθως μάλλον αντιδρά περισσότερο στα προβλήματα που προκύπτουν παρά να προσπαθεί να προλάβει τις κρίσεις όταν προκύπτουν ή να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα βήματα προόδου. Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει αυτό το πρόγραμμα δράσης είναι οι αποτιμήσεις του ευάλωτου χαρακτήρα, κάτι που προκύπτει σε εθνικό, κρατικό επίπεδο. Οι εκθέσεις που ετοιμάζονται οι εκθέσεις που, που ετοιμάζονται δείχνουν πώς οι χώρες ε, αντιλαμβάνονται τον ίδιο τον επανατοχαρακτήρα χαρακτήρα τους και το τι ανάγκες μπορεί να ζητηθεί να καλυφθούν. Θα συνεχίσω την παρουσίαση της μελέτης. αν μπορώ να... Αν μπορώ να, ναι, να χρησιμοποιήσω αυτό το μικρόφωνο. Να κάνω μια σύντομη ιστορική επισκόπηση για το, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εφραυστά κράτη. Το πρόγραμμα για την πρόληψη των βιαίων συγκρούσεων έχουν εδραιώσει την πρόληψη συγκρούσεων ως κύριο πυλώνα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαγάγει την ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία έγινε γνωστή αργότερα ως συνολική προσέγγιση. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 η οποία είχε σαν στόχο την πρόληψη της αστοχίας κρατών μετά από τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου και η συνένεση του 2005 που οδήγησε την Κομισιόν σε μια συνολική αντιμετώπιση της ε, ευθραυστότητας των κρατών και των φυσικών καταστροφών, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2007 για την ανάπτυξη που τόνισαν την σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης, αλλά ακόμα και η εντολή του Συμβουλίου προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ευθραυστότητα και τις συγκρούσεις ο στόχος λοιπόν αυτών των σχεδίων δράσης ήταν να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για το πώς να ενισχύσουμε την ε, απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έθραυστα κράτη με τέσσερις τρόπους. Καταρχήν μια συνολική προσέγγιση, δεύτερον δημιουργία κρατικών δομών, τρίτον να γίνει πιο αποτελεσματική η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτον διεθνείς στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Αυτό που είδαμε όμως ήταν ότι δημιουργήθηκε η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής υπηρεσίες εξωτερικής δράσης, ότι αυτό καθυστέρησε τη δουλειά πάνω στο σχέδιο δράσης. Η ανακοίνωση του 2011 για την ατζέντα αλλαγής έφερε μεγαλύτερη προσοχή στη σύνδεση μεταξύ ανασφάλειας και ένδυας και δέσμευσε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να οριστικοποιήσει και να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης. Το 2012 το Συμβούλιο κατέληξε σε συμπεράσματα για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και ζήτησε από την Κομισιόν και την υπατή εκπρόσωπο να αρθρώσει καλύτερα μια συνολική αντιμετώπιση και πρόσφατα το 2013 η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δημοσίευσαν μια κοινή ανακοίνωση για την συνολική αντιμετώπιση σε εξωτερικές συγκρούσεις. Θα επανέλθω λίγο αργότερα. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπήρξαν πολλές ε, ανησυχίες που αναφέρθηκαν για τον συντονισμό μεταξύ της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και της Κομισιόν, την κατανομή ευθυνών για τα έθραυστα κράτη και τις συγκρούσεις, είναι πράγματι ε, αυτή η ευθύνη μεταξύ της ΔΕΒΚΟ, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των Υπηρεσιών Εξωτερικής Πολιτικής της για κάποιον ο οποίος βρίσκεται έξω από αυτό το κυκαιώνα είναι σχεδόν αδιαφανές πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες και πώς συνδέονται με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική μας κρίση είναι ότι αυτό έχει περιορίσει σημαντικά την αποτελεσματική ανάπτυξη και κατανόηση των διαφόρων εργαλείων που έχουν σαν στόχο να αυξήσουν την αποδοτικότητα σε λειτουργικό επίπεδο. Έρχομαι τώρα στα εργαλεία. Τα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει καταστάσεις συγκρούσεων είναι χωρίς ισοδύναμο σε άλλους χώρους. Έχουμε το DCI, το EMI και το IDHI και έχουμε και βραχυχρόνια εργαλεία όπως είναι το, η διευκόλυνση για την ειρήνη στην Αφρική, η, το εργαλείο για την εξωτερική πολιτική και την ανθρωπιστική υποστήριξη της δημοκρατίας. Και κινητοποιούμε σημαντικά κονδύλια για τη δράση μετά από έκτακτες ανάγκες. Κοιτάξαμε περισσότερο το εργαλείο σταθερότητας, το μέσο σταθερότητας. Η περισσότερη υποστήριξη αυτού του μέσου είναι για χρόνια μη προγραμματιζόμενη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει και μία μακροχρόνια διάσταση που την υποστηρίζει η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση, για δημιουργία κρατικών δομών κτλ. Το, το μέσο σταθερότητα δίνει μονάχα βοήθεια για την πρόληψη συγκρούσεων με την έννοια ότι μια αποτελεσματική απάντηση δεν μπορεί να δοθεί από κανένα άλλο εργαλείο. Είναι περιορισμένη και η χρονική διάρκεια δράσης του 18 με 24 μήνες αλλά αυτό καταδεικνύει ότι και μακροχρονιότερες και προληπτικότερες δράσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενέργειες του DCI. Η χρονικοπεριορισμένη υφή αυτού του εργαλείου επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητά του, γιατί μακροχρονιότερα εργαλεία που προλαμβάνουν συγκρούσεις πολλές φορές δεν μπορούν να καταλήξουν και να οριστικοποιηθούν και έτσι δεν μπορεί να επιτευχθεί μακροχρόνια σταθεροποίηση. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης και τα συμβόλαια για τη δημιουργία κρατικών δομών που είναι σημαντικά εργαλεία για την ε, υποστήριξη του λεγόμενου New Deal για την ε, δημιουργία κρατικών δομών και τη σταθεροποίηση, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα πρακτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν πώς τα συμβόλαια για την οικοδόμηση κρατικών δομών έχουν χρησιμοποιηθεί σε χώρες όπου εφαρμόζεται το New Deal. Κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να λεφτεί για τα συμβόλαια αυτά, για τις συμβάσεις αυτές, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ των εκτιμήσεων ευθραυστότητος του New Deal και των εκτιμήσεων ευθραυστότητος για τα συμβόλαια οικοδόμησης κρατικών δομών, όπου στα τελευταία βλέπουμε να ελείπει η, η παρουσία εταιρικών κυβερνήσεων στη διαδικασία αυτή. Ποια είναι αυτή λοιπόν η συνολική προσέγγιση. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια κοινή κατανόηση της συνολικής αυτής προσέγγισης, η οποία όμως ήταν πάρα πολύ ελληματική και φευγαλαία. Πήρα ένα διάγραμμα από ένα συνάδελφό μας, τον Άντριου Σέριφ, ο οποίος δίνει αυτό το σχηματικό χαρακτήρα σε αυτή τη συνολική προσέγγιση. Γιατί τι θέλουμε πρώτα, ποιος είναι ο στόχος της είναι εργαλείο για την πρόληψη συγκρούσεων, για την αντιμετώπιση των κρίσεων, για την δημιουργία κρατών. Όλα αυτά. Δεύτερον, ποιο και με ποιον εμπλέκεται μέσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ εμπλέκονται τα κρατημέλη, πώ εμπλέκονται οι εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρικανική Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στα Ηνωμένα Έθνη, στην κοινωνία των πολιτών. Πώ λοιπόν που λειτουργεί αυτό, ποιε είναι οι κινητήριε δυνάμει και οι λοκομοτίδες. Πού, το ερώτημα. Πότε. Τι είναι τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα, μακροπρόθεσμα προγράμματα, πώς βγαίνει από ένα τέτοιο σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, πού. Αυτό έχει να κάνει με τη γεωγραφία. Έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση σε τοπικό, ε, περιφερειακό, εθνικό και υπηρετικό επίπεδο. Και πώς συνδέονται αυτές οι διαστάσεις. Επίσης το θέμα του αν θα πρέπει να υπάρχουν γεωγραφικού χαρακτήρα προτεραιότητας ή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έτοιμη να δράσει με τον τρόπο αυτό, με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε ε, ευάλωτο κράτος ή κράτος που έχει να κάνει με συγκρούσεις. Πέμπτον, τι, τι είδους δραστηριότητες στενά στρατιωτικού χαρακτήρα δράσης, ευρύτερες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ασφάλεια, περιλαμβάνει την άμυνα, τη διπλωματία, και την ανάπτυξη ή περιλαμβάνει και το εμπόριο. 6. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Ποιοι είναι οι θεσμικοί μηχανισμοί, ποια είναι η ιεραρχική αλυσίδα ε, για τις αποφάσεις, ποια είναι τα κίνητρα, ποια είναι τα αντικίνητρα. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν θεσπίζει μια σειρά από στόχους δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να έχει μια κοινή ανάλυση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση μια δυνητική κατάσταση κρίση. Επομένω, απαντά στο ερώτημα γιατί. Θέλει να καταλήξει σε μια κοινή στρατηγική ενατένιση οποιασδήποτε κατάσταση σύγκρουση εγκάρση από όλε τι περιοχέ δράση των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Το γιατί και το πού μιλάει για το πώ μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα με του εταίρε μα όπω είναι το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη Κοινωνία των Πολιτών. Το με ποιον ή με ποιαν. Επίση, πώ θα δράσουμε μακροπρόθεσμα ενώ δρούμε και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και εξασφαλίζουμε φυσικέ συνέργειε. Το πότε επομένω αντιμετωπίζει. Επίση, αντιμετωπίζει τα θέματα τη πρόληψη, όταν είναι αυτό δυνατό με διπλωματία και με έγκαιρη προειδοποίηση και με και έγκαιρη δράση. Το τι επομένω και μιλά για το πώς μπορεί να κινητοποιηθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποστήριξη κοινών στόχων. Επομένως το πώς. Και επίσης μιλάει για το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κεντρικό και κωδικό της ρόλο για να υπάρξει συντονισμός του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξουμε κοινό προγραμματισμό με τα κρατημέλη της ενέργειας όλες αυτές. Πάλι ξαναγυρίζουμε στο πώς. Αυτό το οποίο λείπει είναι το πού. δεν λέει πού είναι η γεωγραφική εταιρία, Δεν μας λέει ποιο είναι το σχέδιο δράσης που χρειαζόμαστε. Για το πώς όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν πραγματικότητα και θα πάρουν σάρκα αλλά και ούστα. Προχωρώ τώρα στις αξιολογήσεις που κάναμε. Επί τη βάση της ε, ε, εποπτικής έκθεσης του ΩΣΑ και επί τη βάση και άλλων στοιχείων. Έχουμε και τα θετικά στοιχεία και τα αρνητικά στοιχεία της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταναν στα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής που τονίζει την ανάγκη να υπάρχει μια μακροχρόνια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και είναι σημαντικό, οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τις ρίζες των συγκρούσεων. Αλλά υπάρχει κατακαιρματισμός των ευθυνών γι' αυτό μέσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μια πολύ καλή απόδοση στο να ενθαρρύνει την εγχώρια ικανότητα για να προληφθούν οι συγκρούσεις και έχει υποστηρίξει τις δυνατότητες οικοδόμησης ειρήνης περιφερειακών φορέων μέσω της ε, διευκόλυνσης ειρήνης στην Αφρική και της κοινή ε, δράσης με οργανισμούς όπως το Αζίρ και τα Αλλά δεν έχει επαρκή ικανότητα, αρκετό προσωπικό και εμπειρογνωμοσύνη στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει μια στενή σύνδεση της προσέγγισης ανακούφισης και ανοικοδόμησης, αλλά υπάρχει ένα κενό στην μετάδοση της σκητάλης μεταξύ βραχαίων και μακροπροθεσμών εργαλείων. Το ξεκινήσει λοιπόν μετά από την ανακουφιστική βοήθεια και παρέμβαση η ανοικοδόμηση είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συντονίσει με άλλους εταίρους αλλά η συνεργασία με, το, με τα Ηνωμένα Έθνη παραμένει σε επίπεδο ad hoc. Η συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις έχει παραμείνει σε επίπεδο μονάχα ανταλλαγής πληροφοριών με πολύ λίγα παραδείγματα κοινών στόχων, κοινού προγραμματισμού ή σαφούς κατανομής ρόλων για να ενισχυθούν οι συνέργειες και να αποφευθεί η αλληλοεπικάλυψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει βοήθεια στοχοθετημένα σε μονάχα ορισμένε εύθραυτες περιοχές και περιοχές, αλλά δεν έχει κάνει σημαντική ανάλυση των συγκρούσεων και με ε, μη συνεκτικό και συνεπή τρόπο έχει εξασφαλίσει την χρήση των ε, αξιολογήσεων για την ε, ύπαρξη δυνητικών συγκρούσεων. Το New Deal και η ανάλυση του New Deal μπορεί να είναι ένα σημαντικό παράγον στο να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση των συγκράξεων αυτών και τη ενσωμάτωσή του σε όλο τον προγραμματισμό που σας ενδιαφέρει. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν μια σειρά από προκλήσεις στην αντιμετώπιση των έθραυστων κρατών. Έχουμε κυρίως τι περισσότερε αναλύσει που αφορούν χώρε χαμηλού εισοδήματο. Όπω είπε όμω ο Εδουάρδος, ο συναδέλφό μου, αυτό γίνεται, η εφραυστότητα αφορά και χώρε υψηλότερου εισοδήματο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει αν η αντιμετώπιση τη εφραυστότητα θα πρέπει να καλύπτει μονάχα τα κράτη χαμηλού εισοδήματο, ή αν θα πρέπει να υποστηρίξει περισσότερο την αφεκτικότητα και όχι μονάχα τι χώρε χαμηλού εισοδήματο. Παραδείγματο χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιοχή της Μεσογείου και έχει εμπειρία συνεργασίας με χώρες της περιοχής αυτής που έχουν γνωρίσει την ευθραυστότητα τα κράτη του Κοινοβουλίου. Θα θέλανε να υποστηρίξουν ορισμένου τομεί, ορισμένα θέματα στα κράτη αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν από του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι πολυμερεί ή διμερεί οργανισμοί μπορεί να έχουν περισσότερη εμπειρία και να έχουν και τα κατάλληλα χρήματα. Εμεί θεωρούμε ότι εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή τη είναι στον τομέα της δικαιοσύνης. Εκεί υπάρχουν σημαντικέ προκλήσει για ουσιαστικέ εταιρικέ σχέσει που ξεκινούν από τον πολιτικό τομέα μέχρι την λειτουργικότητα. Υπάρχουν οργανωτικέ συνέπειε που προκύπτουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, τέτοιο, σε τέτοιες ε, εταιρικέ σχέσει, τα θέματα συνεργασία και συντονισμού σε επίπεδο Συμβουλίου υψηλή εκπροσώπου που μετά πρέπει να μεταφραστούν σε στρατηγικέ σε χαμηλότερο επίπεδο στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε επίπεδο των ιδίων αυτών ευθράστων, όσων ευθράστων κρατών και να είναι, με συνεργασία των κρατών μελών. Υπάρχει και η πρόκληση του να μπορέσουν οι αποφάσει Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφράζονται σε συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η ηγέτης του συντονισμού, εκεί θα πρέπει η επικεφαλή των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εμπλεκόμενη στις συζητήσεις αυτές. Εσωτερικός κατακαιρματισμός. Η ευθύνη για τα έφραστα τα κράτη που είναι διάχυτη μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση από το κεντρικό αρχηγείο έναντι τη προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο. Ο συντονισμός που γίνεται μονάχα σε κεντρικό επίπεδο θα κάνει πιο επαχθή και δύσκολη και βαρία και καθυστερημένη την αντιμετώπιση των κινδύνων και την αξιολόγησή τους. Η αποκέντρωση προς την κατεύθυνση των αρχηγών αντιπροσωπιών σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερη εξουσία για το πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι πόροι, αλλά να έχουν και μεγαλύτερη ευκαμψία. Η εμπειρογνωμοσύνη καθώς και η ικανότητα είναι σαφέ ότι οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι διάφορε χώρε αυτέ χρειάζονται τα προσόντα και την σωστή κρίση, την ευθυκρισία να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει επαρκέ προσωπικό και οι επικεφαλεί των αντιπροσωπιών θα πρέπει να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ ψηλό πύχη ώστε να έχουν την επαγγελματική αριστεία για αυτέ τι θέσει. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η μεταβατική περίοδος από το βραχυπρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Τα επιλεγμένα μέσα επιβραδύνουν μερικές φορές την ανάπτυξη των θεσμών, αλλά μερικές φορές καταστρέφουν και ήδη υπάρχουν τα όργανα. Για να ολοκληρώσω. Προτείνουμε, κάνουμε κάποιες συστάσεις. Αλλά πριν φτάσω στις συστάσεις, ίσως θα έπρεπε να τονίσω ότι οι αδυναμίες που φαίνεται να υπάρχουν, που καταδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι διαφορετικές από αυτές που πλήττουν άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Υπάρχει κατακαιρματισμός, Κατακαιρματισμό ε, της πολιτικής ε, δηλαδή μεταξύ διαφορετικών θεσμικών οργάνων, κατακαιρματισμό των πόρων και δεν επενδύουμε αρκετά σε πραγματογνωμοσύνη. Προτείνουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. να ολοκληρώσει το πρόγραμμα δράσης. Είναι ένα σύνολο αρχών. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκρινίσει το ρόλο της και τις ευθύνες της και σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Αυτό αναφέρθηκε και σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν ε, επίσης και κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια. Πρέπει να προχωράμε βήμα-βήμα. Προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε μια ομάδα συντονισμού Κάτι που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, να υπάρχουν δηλαδή τακτικές συναντήσεις τη ΡΕΛΕΞ, όπου να προεδρεύει η υπατή εκπρόσωπο. Συστήνουμε επίσης η εξουσία για αποφάσεις να λαμβάνει υπόψη την ευελιξία. Να έχουν περισσότερε αρμοδιότητε επικεφαλής των αντιπροσωπιών επίση στη νέα διαδικασία προγραμματισμού. Συστήνουμε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει το βάθος της συμμετοχής της και εμπλοκή της στις ασταθείς χώρες. Να δούμε τι γίνεται με την μη ανθρωπιστική βοήθεια και τέλος θα έπρεπε να σκεφτεί ένα διακανονισμό που θα μπαίνουν από κοινού τα κονδύλια και οι πόροι, ακόμα δηλαδή και με πηγές άλλες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέρμαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Μικαέλα. Μου θύμισες ε, το πείμα του Κίπλινγκ που μιλάει για τους ανθρώπους που τα ονόματά τους είναι ποιος, που, πότε, τι. Αυτό μου θύμισες, αυτό το πείμα. Το βρήκα στο ίντερνετ και Γι' αυτό το λέω. Τώρα, μετά τόσα μας είπες, αυτό σχεδιάζω κάπως. Μας έδωσες πολλές πληροφορίες, ανάλυση εκ των έσω. Νομίζω ότι η μεγάλη αξία του τρόπου που αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με διάλογο, με δημοκρατικό διάλογο. Βάζει τους εμπλεκόμενους γύρω από το τραπέζι και τους βάζει να καταλήξουν σε συμβασμό. Και νομίζω ότι αυτή η μέθοδος χρειάζεται εξαγωγή όλο και περισσότερο. Υποτιμούμε τη δικιά μας ικανότητα, τη δυνατότητα που έχουμε να εξάγουμε αυτό το μοντέλο. Το συστήνεις αυτό και για τις ασταθείς χώρες και στην έκθεσή σου το αναφέρεις. Δεύτερον. Συναντήθηκες με επικεφαλής ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών που να διαμαρτύρονταν επειδή θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώριο λιγμών. Γιατί εγώ αυτό έχω αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν. Δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα δεν υπάρχει αρκετό περιθώριο ελιγμόνο. δεν αφήνουν οι Βρυξέλλες δηλαδή τις αντιπροσωπείες να αντιδρούν με ελαστικότητα στις καταστάσεις απέναντι στις οποίες βρίσκονται. Πρέπει να απευθυνθούν στις Βρυξέλλες, οι Βρυξέλλες να έχουν διαβούλευση και έτσι να έχουν απάντηση. Κύριε Σαρτζεντίνη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιχαήλα, ο συνάδελφος Έτουαρτ, νομίζω λέγεστε. Ναι. Είπατε στην αρχή της παρουσίασής σας ότι καλύτερα θα καταφέρουμε στην απάντηση παρά στην πρόληψη. Όντως, θα... αν είχαμε δει τι μας περίμενε, θα μπορούσαμε ίσως να το είχαμε προλάβει μας παρουσιάζει τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν, τα προγράμματα, αλλά αν ήμουν κοινική θα έλεγα ότι αυτό που πραγματικά λείπει με τις ασταθείς χώρες είναι η πολιτική βούληση. Λείπει η επιθυμία να προλαμβάνουμε αντί να αντιμετωπίζουμε κατόπιν ορθής. Χρειάζεται η πολιτική βούληση για αυτή την προσέγγιση, για να μπορούμε να παρεύουμε έγκαιρα. Να, Κεντρική Αφρική. Δεν νομίζω ότι θεωρεί κανεί ότι υπήρχαν ευκαιρίε για σταθερότητα. Παρόλα αυτά, όταν τα πράγματα πήγαν τόσο στραβά όσο πήγανε πρόσφατα, κανένα δεν το περίμενε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα η κυρία Ελένα Ντενίσα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ονομάζομαι Ντενίσα Ελένα Γινέστη και είμαι επικεφαλής της ε, μονάδας για την αντιμετώπιση των ε, κρίσεων. Και είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι επικεφαλής λοιπόν της μονάδας αυτής, του τμήματος αυτού, που φροντίζει για το συντονισμό και την συνοχή των δράσεων της δικιάς μου γενικής διεύθυνσης. Η αποστολή μας είναι ο συντονισμός in-house όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αστάθεια, με την έλλειψη σταθερότητας. Είναι και στο διαδίκτυο της καλλιώς εκθέσεις μας, μπορείτε να τις βρείτε. Έχουμε το πλαίσιο στρατηγικής αποτελεσμάτων, έχουμε την εφαρμογή του New Deal, έχουμε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έχουμε και δομές της ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ και έχουμε επίσης σχέσεις και με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και μεταξύ άλλων προεδρεύω την Διπηρεσιακή Ομάδα για τις Υπηρεσίες. Θέλω να υπογραμμίσω, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται στα δικά μας θεσμικά όργανα τα δύο τελευταία χρόνια. Και αυτό κυρίως γιατί, όπως το είπατε, είναι κάτι πρόσφατο και βασιζόμαστε και σε μια άλλη μελέτη για την πρόληψη των κρίσεων. και την ε, ε, καθίδρυση μιας σταθερής ειρήνης. Από το 2001 μέχρι το 2009 βέβαια γίνανε πολλά. Επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, έχουμε δημοσιεύσει και τον φάκελο με την παρακολούθηση των διαφόρων δράσεων. Θέλω τώρα να μπω στην ουσία της ανάμειξής μας στις ασταθείς χώρες τα τελευταία χρόνια. Από τότε που έχουμε την Agenda for Change και να σας εξηγήσω την κοινή ευρωπαϊκή θέση για το φόρουμ του Μπουσάν που λέει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για μια νέα προσέγγιση απέναντι στις ασταθείς χώρες. Και συγγνώμη βέβαια που ξοδεύω το χρόνο σας κυρίες και κύριοι και κυρία Πρόεδρε, θέλω να αντιδράσω λίγο και σε αυτά που ακούσαμε για το προηγούμενο σημείο και το οποίο φάνηκε και σήμερα το πρωί, γιατί σήμερα το πρωί παρακολούθησα λίγο μέσω του webstream την συζήτηση που κάνατε εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξή. Πρώτον, το state building, η ενίσχυση δηλαδή των κρατικών δομών στις ασταθείς χώρες, σημαίνει και ένα κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στις κρατικές αρχές και τους πολίτες. Γιατί γι' αυτό, γι' αυτούς γίνεται το state building. Το κοινωνικό συμβόλαιο καθορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά των αρχών τοπικών, εθνικών. Ικανότητες, νομιμότητα και δυνατότητα ηγετική. Αυτές ε, τις αρχές τις χρειαζόμαστε. Όμως βλέπουμε σε ασταθείς χώρες να υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Το είπε και Λάκμα νωρίτερα. Από την ε, δημοκρατία του Κονγκό μέχρι δεν ξέρω ποια άλλη χώρα βλέπουμε να μην υπάρχουν τέτοιες δομές. Τώρα την από Γκάνα, Μπουρκίνα Φάσο. Εκεί υπάρχει μια νομιμότητα, υπάρχει ηγεσία. Το κράτος έχει το μονοπόλιο λίγο πολύ της χρήσης βίας. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό υπάρχει και στο διάλογο που κάνουμε με το λεκτικό συνέδριο είναι ότι το state building, η ενίσχυση του κράτους κυρίες και κύριοι, είναι μια πολιτική διαδικασία ενδογενής στο εσωτερικό των χωρών. Εμείς δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε να το τροποποιούμε βάσει της δικιάς μας προοπτικής. Πρέπει να το στηρίξουμε, αναπτύσσοντας τις ικανότητες για να παραμείνει νομιμότητα, να διασφαλίσουμε ότι γίνονται εκλογές που επιτρέπουν μια πολιτική διαδικασία στην οποία να συμμετέχουν όλοι και όχι έξι μήνες μετά από ένα πραξικόπημα, όπως είδαμε στην Κεντρική Αφρική. Τι κάνουμε με την αστυνομία, πώς στηρίζουμε την ασφάλεια στηρίζοντας την ε, αστυνομία. Το κράτος πρέπει να έχει το μονοπόλιο της βίας, αλλά προς όφελος του πολίτη. Δεν πρέπει να επηρεάζουμε εμείς περισσότερο, αλλά πρέπει να στηρίζουμε μια τέτοια διαδικασία με φύ τρόπο, έχοντας κατά νου το κοινωνικό συμβόλαιο. Κατόπιν τούτον, κύριε Πρόεδρε, για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Θέλω να υπογραμμίσω και να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία και κάποιες δράσεις που αναλαμβάνουμε που ελπίζουμε ότι θα μας βάλουν σε καλύτερη θέση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασταθείς αυτές χώρες, να στηρίξουμε την ικανότητα, την νομιμότητα και τον ηγετικό ρόλο του κράτους. Πρώτον, όσον αφορά τους πόρους. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι τα τρία τελευταία χρόνια η δαπάνες στη διμερή βοήθεια για τις ασταθείς χώρες αυξήθηκε προοδευτικά από 45% περίπου το 2010, σήμερα είμαστε στο 55%. Και εδώ δεν προσθέτω και την βοήθεια στην ασφάλεια, στη διατήρηση της ειρήνης και άλλες δράσεις μέσω του African Peace Facility. Συντονισμός, joint programming έχουμε όλο το πλαίσιο ώστε να αρχίσει και πάλι το John Bromley σε διαφορετικές βάσεις από αυτές που είχαμε πριν από λίγο καιρό όταν δεν λειτουργήσε. Ένα λεπτό μου δίνετε. Ε, δεν ξέρω τι να διαλέξω για να σας τα πω σε ένα λεπτό. Λέω μιλήτρια. Κοιτάξτε, μας νοιάζει τόσο πολύ αυτή η ενίσχυση της ικανότητας τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε 12 ε, μέρες κατάρτισης για το προσωπικό μας, για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Εξετάζοντας θέματα ασταθών κρατών, ικανοτήτων και έχουμε ετοιμάσει και μια δοκιμή την οποία θα την χρησιμοποιήσουμε σε μια τέτοια σταθή χώρα και βασιζόμαστε σε μια περιφέρεια σε συνεργασία με άλλους δωρητές. Για το συντονισμό θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς ασχολούμαστε με τον Ιόντολ στη Σομαλία, ότι συμμετέχουμε επίσης στο Τιμολέστε, όπου και εκεί συμμετέχουμε, όπως επίσης και στην Κεντρική Αφρική. Εμείς συνεργαζόμαστε με τους άλλους δωρητές για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι προκλήσεις είναι τρεις. Πρώτον, μην ξεχνάμε, διακόπτη πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρέπει να προχωρήσουμε. Ακούσαμε με τι ενθουσιασμό μας μιλάτε για αυτά τα θέματα και καταλάβαμε πόσο πολύ έχει δουλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά και τα μοντέλα είναι σημαντικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονε μας για τρία λεπτά καθένας παρακαλώ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέρμαν, θέμενη αξία για το διαμεσολαβητικό ρόλο. Απαιτείται μία καλύτερη κατανόηση του τι μπορεί να αποδώσει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι όλα αυτά προφανή, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι απαραίτητο να έχουμε το σωστό πλαίσιο και να καταλάβουμε ότι οι εγχώροι εταίροι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν τη διαδικασία για τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών. Εδώ πράγματι υπάρχει κάποιο έλλειμμα Τώρα έχουμε τους σωστούς ανθρώπους με τις σωστές δεξιότητες που είναι σε θέση να δώσουν μια απάντηση σε επίπεδο κράτους σε αυτές τις ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς. Για την κυρία Σατζεντίνη. Πολιτική θέληση. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την, το ιστορικό και τις, ε, τα ριζικά αίτια της ε, αστάθειας και του των εισμένων κρατών, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και την περιφερειακή διάσταση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αναφερθήκατε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά και το Μάλι είναι μια τέτοια περίπτωση όπου μας κατέλαβε όλους εξ απίνης, αλλά αν λαμβάναμε υπόψη την περιφερειακή διάσταση θα είχαμε κατανοήσει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας επιβεβαιώσω. Αυτά είναι πολύπλοκα θέματα και τα συμβόλαια για την ε, δημιουργία κρατικών δομών μπορούν να είναι πάρα πολύ θετικά για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. Αυτή είναι η εμπειρία που είχαμε, που είδαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο ξέχασα. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα που θέσατε, διάλογος, διαμεσολάβηση, σύμφωνα απόλυτα. Για μας είναι μια, ένα, μια μορφή συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα προς, τα μέσα του 2014 θα εκδώσουμε μια έκθεση που θα λέει αυτό που σας είπα μόλις σε σχέση με τη λεγόμενη ήπια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκπρόσωπο της Κομισιόν θα ήθελα να πω το εξή. Εγώ έβλεπα το έγγραφο κατευθύνσεων που είχε δημοσιεύσει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το πώς αντιμετωπίζουμε την ε, πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης κτλ. Στη σελίδα 15 υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος των ε, υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, την πρόληψη συγκρούσεων, οικοδόμηση ειρήνης. Υπάρχουν πέντε υπηρεσίες στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, άλλες πέντε στην ΤΕΦΚΟ και υπάρχει και το, η μονάδα για το εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Είναι όμως πολύ ασαφές ποιος κάνει τι, ποιος είναι αρμόδιος γιατί, ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος συντονίζει για, την, για τις ε, κατευθύνσεις λοιπόν που αναφέρθηκαν στο σημείο αυτό δεν είμαι σίγουροι ότι υπάρχει μεγάλη σαφήνεια, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ και την κυρία Καβάς και τον κύριο Έντβαρτ που ήρθατε, που μας παρουσιάσατε την ελέτη αυτή. Είναι, μας βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά και μας εμπνέουν για τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ευρωβουλευτές που υπομονητικά βρίσκονται εδώ από σήμερα το πρωί στις 9. Βλέπω ότι τελικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος είναι η βασική ουσία του κοινοβουλίου μας και δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος φεύγει πριν πάρει την απάντηση επειδή ενοχλήθηκε που το εξηγήσαμε ότι ο χρόνος μας περιορίζει. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο σημείο, θα διαχειριστούμε καλά το χρόνο μας τώρα και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για ένα σχέδιο έκθεσης της κυρίας Αργεντίνη. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ξανά την Επιτροπή μας. Τέσσερα χρόνια συνεργαζόμαστε για αυτό το θέμα. Πρόκειται για την πρόθεση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, κυρίως όσον αφορά το ρόλο των εξορρυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρία Σαρτζεντίνη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Λέει η κυρία Σαρτζαντίνη. Και γι' αυτό, γιατί διαπιστώνω ότι κι εγώ καλύτερα μπορώ να συγκεντρωθώ στην γλώσσα μου και γι' αυτό θα μιλήσω Ολλανδικά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Συνεπώς, ελπίζω να είμαι σύντομη. Θέλω να σας πω ότι φυσικά βρίσκω και εγώ πολύ κρίμα που είναι τόσο λίγοι οι παρόντες συνάδελφοι, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ εσάς που παραμένετε στην αίθουσα και μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Περιμένω να μου κάνετε σχόλια, ό,τι τροπολογίες θέλετε κτλ. Είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, για μένα πρόκειται για μια έκθεση που αναφέρεται στην ε, ανάπτυξη σε σχέση με τις πρακτικές των εξορρυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι ο τίτλος εξάλλου της έκθεσης αυτής, μεγάλος τίτλος, τι να κάνουμε. Μια τέτοια έκθεση πάντως για μένα λέει πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε στις αναπτυσσόμενες χώρες να βοηθήσουμε με καλές πρακτικές από τις εξωτερικές βιομηχανίες και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συνοχή στην πολιτική που ακολουθούμε. Η Επιτροπή μας αυτή ανάπτυξης νομίζω ότι έτσι καλώς ασχολείται με την αναπτυξιακή βοήθεια, πολύ καλό, αλλά επιπλέον πρέπει να ασχοληθεί και με την συνοχή της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής. Στην επαγγελματική μου ζωή 13 χρόνια ασχολήθηκα με έρευνα στα ορυκτά και την ανάπτυξη. Και πριν από 13 χρόνια είχα μιλήσει με την κυβέρνηση της Μποτσουάνα και είχαν θυμώσει τότε. Πρόκειται για τα διαμάντια και την ιστορία αυτή, τα διαμάντια τα βαμμένα μέμα, όπως τα λέγαμε, είχε να κάνει και με τη Σιέρα Λεώνα και με την Αγκόλα και το Κονγκό. Και μετά καταλήξαμε στα διαμάντια για την ανάπτυξη. Ισχύει. Η έκθεση αυτή ακριβώς αυτό θέλει να καταδείξει. Πώς πρέπει να οργανωθεί η εξόριξη ορυκτών σε αναπτυσσόμενες χώρες για να βοηθούν στην ανάπτυξη. Ψηφίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές Χτες ή προχτές η Επιτροπή Γιούρη ασχολήθηκε με την ε, μη δημοσιονομική πτυχή. Τώρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψουμε ώστε οι επιχειρήσεις με διαφάνεια να προχωρούν στις εξοριστικές τους δραστηριότητες. Πιστεύω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι η αναπτυξιακή μας βοήθεια, αλλά και οι υπορικέ μας πρακτικές να είναι τέτοιες που να συνάδουν με την πραγματική ανάπτυξη. Περί αυτού πρόκειται αυτή η έκθεση. Πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση και πώς θα φροντίσουμε να λειτουργήσει καλά η δικιά μας Ήμουν στο Δυτικό Κονγκό πριν από λίγο καιρό, σε ορυχεία κασίτερου μεταξύ άλλων, και εκεί είδα πώς γίνεται η εξόριξη και πώς καταλήγει στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να... Και είδα συγχρόνω πώ γίνεται με του φόρου, πώ πληρώνονται οι φόροι, πώ μπορεί να αποφεληθεί ο ντόπιο πληθυσμό από την εξόριξη αυτή. Ο τόπιο πληθυσμό όμω ήταν θυμωμένο. Είπαν ότι τελικά όλε αυτέ οι ρυθμίσει δεν λειτουργούν, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει δεν κάνουν αυτό που πρέπει και ότι από τότε που έχουν αναμειχθεί οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, κερδίζουμε λιγότερα, ενώ όταν υπήρχε το λαθρεμπόριο κερδίζαμε περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Λίγοι είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Πρέπει να δούμε λοιπόν την εξωστική δραστηριότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Να δούμε επίσης το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Τι μπορεί να κάνει καλύτερα επιτόπου. Πρέπει να δούμε επίσης τα καθεστώτα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων που παραμένει ένα πολύ βασικό θέμα. Η εξαγωγή και η εισαγωγή πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πότε είναι πιο φτηνή και πώς πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Πρέπει να υποφεληθούμε, να φροντίσουμε μάλλον ο ντόπιος πληθυσμό να υποφελείται από τα έσοδα από την εξόριξη ορεκτών και τα χρήματα να μην πηγαίνουν πάντα στην πρωτεύουσα, αλλά να μένουν στα χέρια του ντόπιου πληθυσμού εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα ορυχεία. Πώς λοιπόν θα το πετύχουμε αυτό, πώς δεν θα φύγουν τα χρήματα και δεν θα καταλήγουν αλλού. Αλλά θα κερδίζει και ο ντόπιο πληθυσμό ε, χρήματα από αυτή τη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θέτει και το θέμα των σειράξεων και τη σχέση της εξόρυξης χρυσού και κασίτερου με τις σειράξεις. Δυστυχώς αναβλήθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα με την Επιτροπή. Είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου Τεγούφτ. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να περιμένουμε ακόμα. Πάντως το σημαντικό είναι στη δικιά μου την έκθεση να δούμε την οπτική γωνία της Αναπτυξιακής Επιτροπής και να φροντίσουμε να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να μην ασχοληθούμε μόνο με τις ρυθμίσεις για τις εισαγωγές αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει, να προτείνει ρυθμίσεις όπως τις έχει ανακοινώσει για την βιώσιμη ανάπτυξη εκεί όπου υπάρχουν σειράξεις που απορρέουν από την εξόριξη μεταλλευμάτων. Εκεί πρέπει να δούμε τι μέτρα θα λάβουμε. Κύριε Πρόεδρε, και ζητάω βοήθεια και από εσά και από την Γραμματεία για την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Γιατί δεν το ξέρω αυτό ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Περιμένω να μου πείτε. Ευχαριστώ. Να απαντήσω αμέσως στην ερώτηση της κυρίας Σαρχεντίνη. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Ιανουαρίου το μεσημέρι και ψηφοφορία στις 21 Ιανουαρίου. Τώρα ο λόγος στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτζεντίνη. Ο σκιώδης εισηγητής μας δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την θαυμάσια εργασία της κυρίας Σαρτζεντίνη για το θέμα αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα αυτά που λέει, είναι πολύ καλή η έκθεσή της. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στη συνέχεια σε μερικά σχόλια στις ε, ιδέες που θεωρεί η σοσιαλιστική ομάδα ότι μπορούν να προσθετούν σε αυτή την έκθεση. Υπάρχει ένας κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαφάνεια και ευθύνη στη χρήση των φυσικών πόρων επί τη βάση των ε, προδιαγραφών του ΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών και αυτά είναι όλα αυτά που έχουν γίνει δεκτά σε σχέση με, την, ε, με το θεματολόγιο του 2015. Και υπάρχει αυτή η θέληση να υπάρχει μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την ατζέντα που θα ακολουθήσει το 2015. Αλλά η Κομισιόν με επικεφαλή στον Επίτροπο Χούχτ αναρωτιέται πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό του εμπορίου και της ε, αγοραπολισίας με υπεύθυνο τρόπο των ορυκτών αυτών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεώσει για τι επιχείρησει που λειτουργούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν οι οποίε εξορίσουν τους ε, φυσικούς πόρους και θα πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε όλη την αλυσίδα παραγωγή στηρούνται οι προδιαγραφέ του ΩΣΑ. Θα πρέπει να καταδεικνύεται ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από τις επιχειρήσεις ότι με τον τρόπο αυτό δεν χρηματοδοτούν την κατάχρηση και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και ήθελα από στην κυρία Σατζεντίνη όχι εξ του κυρίου Κάσμαν, αλλά και από δική μου άποψη, εγώ είχα πάει στην Τανζανία να δω ποια είναι η κατάσταση για τις εξορρυκτικές ε, επιχειρήσεις, κυρίως ευρωπαϊκές, στην Ουγγάντα και στην Τανζανία και η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι εύκολο να το διερευνήσει κανεί αυτό. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε τα θέματα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν αφορά μόνο την Αφρική. Και σε άλλε περιοχέ, στη Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν ε, εξορυκτικέ ενέργειε, υπάρχουν σημαντικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και είναι κρίμα που δεν υπάρχουν ε, περισσότεροι βουλευτέ για να μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα αυτά που νομίζω ότι επέχει τεράστια σημασία. Και απλώς θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια ότι έχει την απόλυτη υποστήριξή μας για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα φιλόδοξο έργο, σε μια φιλόδοξη έκθεση της οποίας ο κύριος στόχος θα είναι να μπορέσουν να σταματήσουν ορισμένες καταχρήσεις οι οποίες γίνονται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εξοριστικές εταιρείες στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λεβίν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που και εγώ μπορώ να μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Κάτοτε που είναι πάντοτε ευχάριστο. Είναι λίγοι συνάδελφοι, οπότε θα λάβω και εγώ το λόγο για να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γιούντιτ για την ε, άρτια και διεξοδική έκθεση που συνέταξε. Όπως είπε ο κύριος Κόρτες Λάστρα, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να είμαστε υπεύθυνοι στη στάση μας όταν πρόκειται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με ορυχεία, με εξορυχτικέ βιομηχανίε, με μεταλλεύματα. Ιδίω σε τρίτε χώρε. Υπάρχει μια σειρά από καλέ προτάσει στην έκθεση τη Judith και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε εξορρυκτικές εταιρείε να πληρώνουν φόρου στι ε, χώρε. χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Το να υπάρχουν φορολογικέ συμφωνίε με τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ε, αντικείμενο διαπραγματεύσεων, όπω σωστά επισημαίνει στο σημείο 26 η Judith. Πολύ καλή ιδέα. Η, η η, η δυνατότητα ανείχνευση των ε, μεταλλευμάτων, ώστε να βρεθεί ποια ήταν η προέλευσή του εφόσον χρειαστεί, είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να το αναλάβουμε ω ευθύνη. Διάβασα την έκθεση, κάπως βιαστικά βέβαια, αλλά διερωτώ με αν κάπου γίνεται λόγος για την ε, πρωτοβουλία διαφάνειας της εξωτερικής βιομηχανίας, δηλαδή αν θα δημοσιεύονται αυτά που πληρώνουν. Μήπως λοιπόν αν δεν υπάρχει αυτό στην έκθεση θα πρέπει κάτι να προσθέσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, οπότε γι' αυτό θα μιλήσω και εγώ τη δική μου μητρική γλώσσα. Τα νορβηγικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Σαρχιντίνη, για την εξαιρετική σας έκθεση. Πολύ σημαντική. Νομίζω ότι περατώνεται αισίως αυτό που επιδιώκαμε εδώ και 4,5 χρόνια. Και εδώ έχουμε μια πραγματική ένδειξη για το πραγματικό περιεχόμενο της βοήθειας. Δεν είναι μόνο χρήματα ή ποσά βοήθειας δεν είναι μόνο το 7,7 το 0 μάλλον κόμμα 0,7 ε, του ΑΕΠ που θα πρέπει να συγκεντρώνεται. Η βοήθεια έχει να κάνει με τα φορολογικά συστήματα, τους φορολογικούς παραδείσους, όπως σωστά τους εντοπίζει η κυρία Σαρχεντίνη στην παράγραφο 27. Νομίζω ότι η παράγραφος 20 είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί λέτε εκεί ότι για μας είναι σημαντικό να έχουμε διαρκώς κατά νου ότι έχουμε προσφέρει πολλά, ε, πολύ μεγάλα ποσά στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν ξέρουμε πού καταλήξαν τελικά. Ε, λόγου χάρη βλέπουμε πόσο έχει εξαπλωθεί η Γερμανία στον υπόλοιπο κόσμο και ξέρουμε τι έγινε στο Μάλι, όπου οι εξορρυκτικές μηχανίες δεν κατέβαλαν κανένα φόρο, δεν ανέλαβαν ένα μερίδιο ευθύνη στην οικονομία της χώρας. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για καναδέζικες εταιρείε. Δεν πληρώνουν όταν δραστηριοποιούνται σε τέτοιες χώρες. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η έκθεση αυτή εκπροσωπεί την πεμπτουσία του έργου αυτής της Επιτροπής. Νομίζω μάλιστα ότι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις προέκυψε συνένεση ως προς την θέση αυτή. τη θέση αυτή για την αναπτυξιακή πολιτική. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ την κυρία Σαρχεντίνη για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την σκληρή προσπάθειά τους να πετύχουν την νορβηγική μου προφορά. Δεν είναι ακριβώ σουηδικά, μοιάζουν. Πάντως ήταν μεγάλη μου χαρά σε αυτή την τελευταία συνεδρία πριν τα Χριστούγεννα να εκφραστώ στην γλώσσα μου. Τώρα στα 5 ή 6 λεπτά που μας μένουν να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην αισθανθείτε όμω προσβεβλημένοι αν σας διακόψω γιατί εξαντλήθηκε ο χρόνος σας. Ο κύριος Κόρτζη και ο κύριος Νίλαντ. Μπορείτε να λάβετε το λόγο. Με όποια σειρά θέλετε. 5 με 6 λεπτά και οι δύο. Παρακαλώ. Um, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Δεν θα χρησιμοποιήσω όλα στις σημειώσεις 22 σελίδες που μου δώσανε για αυτή την ε, ενημέρωση. Αυτό είναι ένα άλλο αρνητικό στοιχείο της ε, έλλειψης χρόνου. Έχω συμμετάσχει τουλάχιστον σε τρεις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την εξόριξη φυσικών πόρων τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό και κατεπήγον θέμα. Είμαι στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Αν θέλετε λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την οπτική γωνία της ανάπτυξης προτού δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου της Digitrade. Νομίζω ότι γενικά μπορούμε και εμείς να συγχαρούμε την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνούμε στα περισσότερα σημεία αυτής της έκθεσης και συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας. Πάντα βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία όπου η Κομισιόν θα έχει ακολουθήσει μία διαφορετική διατύπωση. Ανθρώπινο είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της παρέμβασής μου. Πιστεύουμε ότι αν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο η έκθεση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί, θα μπορούσε να είναι να δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία και ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με ορισμένε δηλώσεις που κάνει η συγγητρία. Τονίζω και πάλι ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο σε μεγάλο βαθμό, αλλά το να υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις και ποσοτικοποίηση <clears throat> θα ενίσχυε και το έργο της έκθεσης. Η κλίμαξ, παραδείγματος χάρη και τα διάφορα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί εάν δεν αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι συμφωνούμε ότι πρέπει να αναλυθεί δράση σε πολλές περιπτώσεις και το έχουμε κάνει. Αλλά θα έπρεπε να αξιολογήσουμε και τις δύο δυνατότητες δράση ή μη δράση. Τουλάχιστον συστηματικού χαρακτήρα. Και υπάρχει μετά το θέμα τη αποτελεσματικότητα και τη αναλογικότητα των δράσεων που προτείνονται από την έκθεση τη κυρία Γεντίνη. Αυτά εν συνοπτικότητο, εν συνοπτικότητη τα σχόλιά μου και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε μια άλλη ευκαιρία την συζήτηση αυτή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω τα διαφορετικά στοιχεία που κατά τη δική μας άποψη είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί το βασικό θέμα του πώς να μεταμορφώσουμε την, ε, το δυναμικό που υπάρχει για την εξόρυξη σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Δεν έχουμε παρουσιάσει κάτι το οποίο είναι <clears throat> ριζικά διαφορετικό. Το έχουμε τονίσει σε διάφορες συναντήσεις και ενώπιον της δικής σας Επιτροπής. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε καλύτερη γνώση των πόρων, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα ήταν σε καλύτερη θέση αν ξέραν καλύτερα τι φυσικούς πόρους διαθέτουν. Επίσης, να απαραίτητη η ικανότητα να κάνουν πραγματικές και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις. Μια αποτελεσματική φορολογική πολιτική, διαφάνεια, καλύτερος ρόλος του επιχειρηματικού πλαισίου και του ιδιωτικού τομέα και τέλος καλύτερη γνώση για το πώς να υπάρξει αηφόρος εκμετάλλευση των φυσικών πόρων η περιβαλλοντική πλευρά. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο σε αυτά, γιατί όπως σας είπα τα έχουμε συζητήσει σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες ευκαιρίες. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους μου να καλύψουν και την πτυχή του εμπορίου που την ανέφερε η εισηγητρία. Αμέσως θα συνεχίσω. Νίλαντ από την GG Trade Εργαζόμαστε τον τελευταίο χρόνο για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές σύγκρουσης. Θέλω να συμμεριστώ ορισμένα σχόλια που ίσως ενδυναμώσουν αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι στα τελευταία τμήματα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και αυτά που λέγονται στην, ε, στο νομο dodge Dodd-Frank. Εκεί υπάρχει ήδη μια δύναμη η οποία σπρώχνει τις αμερικανικές εταιρείες προς την κατεύθυνση αυτή. Αν το λάβουμε αυτό υπόψη, θα μας καταδείξει και ποια είναι τα προβλήματα που έχουν αυτές οι, οι εταιρείε. Υπάρχει μια πίεση που ασκείται στις ευρωπαϊκές εταιρείε γιατί είναι πολύ μακρά η αλυσίδα παραγωγής και μεταφοράς για τα ορυκτά. Ε, όταν λέει η έκθεση ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το ανάντι και το κατάντι το ανάντι υπόκειται στην ε, νομοθεσία Dodd-Frank, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλες αυτές οι απαιτήσει. Θα πρέπει επομένως εμείς να βοηθήσουμε αυτές τις εταιρείε. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση στο τμήμα που είναι ανάντι και όχι στο τμήμα που είναι κατάντι. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ενσωματώσουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την νομοθεσία Dodd-Frank είναι η απόσταση των επιχειρήσεων από τις περιφέρειες όπου δρούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται στην έκθεση, αλλά είναι <clears throat> κάτι όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διδαχθεί και βλέπω και το ορολόγιο. Αυτό λοιπόν θα ενίσχυε, και αυτό είναι το τελικό μου σχόλιο, θα ενίσχυε και την έκθεση. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο και ξαναδίνω τώρα το λόγο στην εισηγήτριά μας για πέντε λεπτά για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και στα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις φιλοφρονήσεις τους. Είναι πάντοτε ευχάριστες. Να πω το εξή για αυτή την έκθεση. Γιατί να μην είμαστε όλοι σαν την Νορβηγία. Γιατί τα εμπορεύματά μας να μην τα χρησιμοποιούμε με τρόπο υπεύθυνο, να τα χειριζόμαστε με μια διορατικότητα για το μέλλον. Γιατί να μην είμαστε όλοι Νορβηγία ή γιατί να μην είμαστε όλοι σαν την Ποτσουάνα που έχει μια ευφυή διαχείριση του θέματος των αδαμαντορυχίων. Το θέμα λοιπόν με, την, με τους φυσικούς πόρους είναι μια διελκυστίνδα διαρκή είναι σαν την κότα με το αυγό. Δηλαδή οι εταιρείε είναι εκεί γιατί υπάρχουν οι πόροι ή το αντίστροφο. Κανεί δεν θα βρει ποτέ την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Όμω μπορούμε να βρούμε και να σχεδιάσουμε πολιτικέ λύσει που να βελτιώνουν τα πράγματα. Φτάνοντα στην ερώτηση τη κυρία Λέβιν. Ναι, υπάρχουν αναφορές στο τι πρέπει να καταβάλει η κάθε εξωτερική εταιρεία με αφορμή την έκθεση της Transparency International. Ε, πολύ σωστά δημοσιεύτηκε η έκθεση αυτή. Εγώ ήμουν εκεί στην πρώτη της ε, δημοσίευση, αλλά μιλούσα πιο πολύ για ε, εθελοντικά προγράμματα, τα οποία τελικά απαιτούν νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού. Ένα παράδειγμα, το γεγονός ότι το Κονγκό, η Αγγόλα και το Τσάντ ακόμη δεν είναι μέρος του του ITI δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα. Ακόμη και η Νότιος Αφρική και όσοι πήγαν στην αποστολή στην Νότια Αφρική δεν έχουν συγκληθεί στην ε, διεθνή αυτή συνθήκη. Οπότε πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη νομοθεσία ώστε να επιβάλλεται η εταιρική ευθύνη και όχι μόνο εθελοντικά προγράμματα. Αυτό επιδιώκω ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να έχετε διάθεση να μας δώσετε και εμάς τις 22 σελίδες κειμένου που έχετε ώστε εγώ και η Συμβουλή μου να διαφωτιστούμε και να καταλάβουμε ακριβώς πού χρειάζεστε περισσότερα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα. Διότι προφανώς, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε αυτό το νομοθέτημα να το βελτιώσουμε, ε, θα δεχτώ κάθε βοήθεια. Εάν λοιπόν έχετε συγκεκριμένα σημεία όπου χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις, μακάρι να μας τις προσφέρετε. Στον κύριο Νίλαντ της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, ναι, συζητήσαμε γι' αυτό και στο παρελθόν και γνωρίζω πολύ καλά ότι το ρεύμα στο δωμάτιο ε, είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα θέλα να αλλάξει. Δηλαδή, από το Ανατολικό Κονγκό η ροή καταλήγει με την διαχείριση των φυσικών πόρων που έχουμε εκεί στην ανάγκη για ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή η Κινσάσα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα των ορυχείων και έχει γκρίζα και κόκκινα ορυχεία και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα πιο διαφανή και προσπαθεί να ε, εξηγιάνει τον εξορρυκτικό τομέα. Αυτό είναι ευχάριστο όμως δεν λειτουργεί ακόμη ε, το σύστημα. Οι εταιρείε φεύγουν. Το εξορισμό εμπάργκο πρέπει να διαραγεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα θέματα ε, κατάντι, αλλά και ανάντι, να δημιουργηθεί μια νέα αγορά για προϊόντα που δεν έχουν σχέση με ε, σύραξη. Δηλαδή ε, ανιχνεύσιμα μεταλλεύματα ή προϊόντα μεταλλευμάτων. Ελπίζω ότι η πρότασή σας στην Άνοιξη να μην αντιμετωπίζει μόνο την ανάντι διάσταση, αλλά και την νομοθεσία που εμείς οφείλουμε να ε, έχουμε στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, διότι το Dodd Φράγκ δεν θα το βελτιώσουμε εάν δεν υπάρξει κάτι από τα δύο νομοθετήματα που χρειάζονται. Θα ήθελα λοιπόν να μας κάνετε μια πρόταση που να δώσει στην εταιρεία αυτή τη ε, δυνατότητα να επακούσει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα και στην Αμερικανική. Τέλο πάντων, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η έκκλησή μου προ εσά. είναι η έκκλησή μου προ τον Επίτροπο που ακούει αυτή την έκκληση εδώ και καιρό και εδώ θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Διορθώνω αυτό που είπα, η προθεσμία για τι τροπολογίες είναι 16 Ιανουαρίου το μεσημέρι, η ψηφοφορία στι 11 Φεβρουαρίου και όχι 21 Ιανουαρίου όπω λαθασμένα είπα. Εάν δεν υπάρχουν διάφορα, μπορώ να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες στις 20 Ιανουαρίου από τις 15, 18 και 30 και την Τρίτη 21 από τις 9 ως τις 12.30 και από τις 15 ως 18 και 30. Σας ευχαριστώ όλους εκ βάθους και σας εύχομαι καλές γιορτές.